Liebe Kolleginnen Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος μετά τις ε, θερινές διακοπές. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε και να επανήλθατε γεμάτη ενέργεια για το φιλόδοξο πρόγραμμα που πρέπει να ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ήδη την πρώτη εβδομάδα συνεδριάσεων έχουμε συνεδρίαση πέμπτη απόγευμα. Αυτό είναι λίγο περίεργο, αλλά έχουμε παρτία και μπορούμε να ξεκινήσουμε με την εξέταση της ημερήσιας διάταξης. Πρώτο σημείο, δεν υπάρχει καμία επιθυμία για τροποποίηση, οπότε ε, έλυσε το θέμα αυτό. Δεύτερον, ανακοινώσεις δικές μου. Δύο έχουν γίνει. Ο Γιώργος Χατζημαρκάκης ε, θα αντικατασταθεί από την Μπρίτα Ράιμερς και ο Τζον Μαρία Ούτσες θα αντικατασταθεί από τον Ανδρέα Τσανόνη. Καλώς ήρθατε νέοι συνάδελφοι στην Επιτροπή μας. την επόμενη φορά θα έρθει εδώ ο αντικαταστάτης σας, ωραία. Στις 31 Αυγούστου Είχαμε την ε, παρουσίαση της αξιολόγησης ε, του προγράμματος περιβάλλοντος από πλευράς της Επιτροπής. Ε, θα εκπονήσουμε έκθεση πρωτοβουλίας υπό το φως και, και του εβδόμου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, διότι το έκτο λύγει τον Ιούλιο του 2012. Θέλουμε λοιπόν ένα έβδομο πρόγραμμα δράσης. Σήμερα, στη Νότια Αφρική, ε, στο Ιωάννεσπουργκ πραγματοποιείται συνάντηση για προετοιμασία της επόμενης διάσκεψης για το κλίμα στο Ντέρβαν. Ήδη ε, έγινε συνάντηση των ε, ανεπτυσσόμενων χωρών, των χωρών basic, που, των αναδυόμενων οικονομιών, που ε, επιθυμούν ένα δεύτερο πρωτόκολλο του Κιώτο. Εμείς ε, έχουμε... Ε, επίσης υπάρχει ένα, ένα αίτημα από την Αυστρία για εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας. Και, και ε, επίσης ε, έχουμε τις ε, προσπάθειες για μείωση της σπατάλης του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης έχουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αυτή τη βδομάδα για το μέλι και τη μόλυνση του από γενικά τροποποιημένους οργανισμούς. Το δικαστήριο πήρε το μέρος των, των παραγωγών ε, μελιού. Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση που θα έχει πολλές ε, συνέπειες. Ε, και όσον αφορά τους γεννητικά τροποποιημένους οργανισμούς στην Ευρώπη. Σίγουρα χρειάζονται μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των καλλιεργιών, διότι οι μέλισσε ε, μπορούν να πετάξουν ακόμα και 16 χιλιόμετρα μακριά. Επίσης, ε, να ε, αναφερθώ σε δύο σεμινάρια που θα γίνουν. Η Ομάδα Εργασίας για την Υγεία στις 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσει σεμινάριο για το θέμα της επιληψίας. Της ασθένειας αυτής που πλήττει αρκετά εκατομμύρια ανθρώπου ε, στην Ευρώπη και επίσης ε, ένα σεμινάριο για την εναλλακτική γιατρική. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις για πράγματα που έγιναν μέσα στο καλοκαίρι, εάν συμφωνείτε. Και επειδή έχουμε πολύ γεμάτο πρόγραμμα, προχωράμε αμέσως στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2012. Όλα τα τμήματα. Ε, Συντάκτη της νομοδότησης είναι η Utah Hawk. Έχουμε μια σειρά τροπολογιών, ε, τις οποίες θα πρέπει να ψηφίσουμε. Προχωράμε λοιπόν κατευθείαν ε, στην ψηφοφορία, εκτός αν η συγγήτρια θέλει το λόγο. Λίγες ε, μονάχα ενδείξεις θέλω να σας δείσω. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι δεν ψηφίσουμε τώρα για το οριστικό για την οριστική θέση. Είχα επαφές με τους σκιώδεις εισηγητές ε, την προηγούμενη Τρίτη. Τους εξήγησα και πάλι ποιες ήταν οι προτάσεις μου για την ψηφοφορία και προσπάθησα να τις ε, αιτιολογήσω κιόλα. Για το ψήφισμά μας τώρα θα ήθελα να πω το εξή. Εγώ προσπάθησα να τα παρουσιάσω όλα με ένα τρόπο ο οποίος να είναι πραγματικά λογικός. Και γιατί να είναι κανείς εναντίον αυτών. Παραδείγματο χάρη αναφέρομαι στο ψήφισμα του, στην τροπολογία του κ. Σκυλακάκη. Δεν μπορούμε να τα καταγράψουμε όλα επακριβώς για τον προϋπολογισμό του 2012. Εμείς έχουμε κρατήσει μια θετική στάση ως Κοινοβούλιο τρεις φορές στο παρελθόν σε σχέση με την στρατηγική Ευρώπη 2020. Επομένως, ακριβώς εκεί που δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, εγώ δεν μπορώ να σταθώ εναντίον. Δεν θέλω λοιπόν να προσπαθήσω να τα βάλω όλα μέσα σε ένα ψήφισμα που αφορά μονάχα το 2012, ένα χρόνο δηλαδή. Επίσης, για αυτό το οποίο ζήτησε η Κορίν Λεπάζ. Ήθελε ή θέλει ακόμα κατά πασαφθανότητα να τεθεί ένα 5% των κονδυλίων της ε, τροφιμικής αρχής της ΕΦΣΑ στο αποθεματικό λόγω του γεγονότος ότι θεωρεί ότι δεν έχουν επιληθεί ακόμα τα προβλήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Δεν έχει εδρεωθεί ακόμα η διαδικασία για τα θέματα αυτά. Συμφωνώ σε αυτό. <clears throat> Και εγώ είδα στην ε, ε, ΕΦΣΑ πόσες προσπάθειες κατέβαλε για να επιλύσει τα προβλήματα αυτά. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση κατά κάποιο τρόπο. Αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον ως αρμόδια επιτροπή προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι συνομιλητές μου στην ΕΦΣΑ προσπάθησαν να με αποτρέψουν στο να υπάρξει μια μεμονωμένη εξέταση τεσσάρων μονάχα αποκεντρωμένων φορέων για τον τρόπο με τον οποίο έχουν αντιμετωπίσει τη σύγκρουση ε, συμφερόντων. Μπορούμε πάντα να εξασφαλίσουμε ότι η ΕΦΣΑ θα τηρήσει αυτή τη διαδικασία για την ε, αντιμετώπιση των σύγκρουσεων συμφερόντων, αλλά αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε κυρώσει εναντίον Το τελευταίο μου σχόλιο. Εφέτος δεν έχω δώσει κανένα, καμία πρόταση για τα προπαρασκευαστικά μέτρα και τα πιλωτικά προγράμματα. Το έκανα σαφέ και στου σκιώδει συζητητέ Πέρσι, <clears throat> κάναμε πολλέ προσπάθειε οι συνεργάτες μου η Κάτια και εγώ ίδια για τα πιλωτικά προγράμματα προσπαθήσαμε να συλλέξουμε όλες τις ιδέες οι οποίες προτάθηκαν από τους συναδέλφους προσπαθήσαμε να τις διασταυρώσουμε να δούμε αν όλα αυτά τα πράγματα τα οποία προτείνονται υπάρχουν ήδη και κατά πόσο μπορούν όλα αυτά να καλυφθούν οι αξίες, να καλυφθούν από πιλωτικά προγράμματα. Δαπανίσαμε ώρες και ώρες για να φτιάξουμε ένα σχέδιο για τα πιλωτικά προγράμματα. Στο τέλος, όταν ήρθαμε στην ψηφοφορία, είπανε τα πολιτικά κόμματα με κάποιο αφαίρετο τρόπο αποφάσισαν να ψηφίσουν. Δεν λάβανε καθόλου υπόψη τις προτάσεις, τις τεκμηριωμένες που είχαμε υποβάλει και επομένω η στάση τη Επιτροπή Προπολογισμών ήταν ουσιαστικά απόλυτα αρνητική. Γι' αυτό εγώ εφέτο δεν κάνω καμιά αξιολόγηση. Απλώ σα ζητώ να κοιτάξει κανεί τι έχει προτείνει η Κομισιόν, τι έχει αξιολογήσει σε σχέση με τέτοιου είδου ενέργειε. Και έχω ζητήσει μετά από τι ομάδε πολιτικέ να προσπαθήσουν να συμφωνήσουν μεταξύ τους για μια ιεράρχηση όλων αυτών των προτεραιοτήτων και η οποία στη συνέχεια θα υποστηριχθεί από τα κόμματα αυτά στην Επιτροπή Προπολογισμών. Όλα τα άλλα είναι στη διακριτική ευχαίρεια τη Επιτροπή μα. Εντάξει, Γιούτα, η σοφία και η σοφροσύνη τη Επιτροπή μα θα φανεί τώρα στην ψηφοφορία την οποία ξεκινάμε. <clears throat> Έχουμε την τροπολογία 600 πρώτα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. κατά. δεκτή. 6301 υπέρ. Κατά. Αποχέ. δεκτή. 17.01.01 με προφορική τροποποίηση ήτριας υπέρ κατά αποχές δεκτή. 63.03 της Κορίν Λεπάζ υπέρ κατά αποχές απολύτω. 63.05 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6302 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6306 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6307 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6308 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6309 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6310 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6338 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6311 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή. 63-12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 63-13 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή. 63-14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 63-15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6316 16 υπέρ και, συγγνώμη, 63-37 υπέρ, είναι ταυτόσιμες, κατά, αποχές δεκτες 6317 63-17 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις Δεν υπάρχουν σχόλια της συζήτησης, όμως στην 63-33. Κατά. Αποχές δεκτή. 63-19. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 63-20. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 63-21. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 63-22 υπέρ κατά αποχές θέλουμε έλεγχο άρχεται η ψηφοφορία πέρας 27 υπέρ 20 κατά καθόλου αποχές εγκρίνεται επομένως 6325 Παναγιώτοφ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6326 υπέρ υπέρ κατά αποχές δεκτή 6327 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6328 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6329 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6332 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6335 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6336 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 63 40 υπέρ κατά απόχες δεκτή 63 41 υπέρ κατά απόχες δεκτή 63 39 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 63-34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε. 63-34. Άρχεται ο έλεγχος. Πέρας. Ναι, ήταν σαφές. 28-19. 63-42. Υπέρ. Κατά αποχές 6318 63-18 υπέρ κατά αποχές 6323 63-23 υπέρ κατά αποχές 6304 63-04 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63-31 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Πέρας προφορίας. Δεκτή. 63-24. Ούλμερ, υπέρ. Κατά. Άποχες δεκτή. 63-30, υπέρ. Κατά. Άποχες δεκτή. Αυτές ήταν οι τροπολογίες επί του προϋπολογισμού. Ερχόμαστε τώρα στο ψ, ψήφισμα για το σχέδιο προϋπολογισμού 2012 ως τροποποιηθέν από το Συμβούλιο. Τροπολογία 1. Ψήφι Dagegen. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Έχει μπλοκάρει το μηχάνημα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2, τη ψηφοφορία, πρώτο μέρος. Υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές ένας υπέρ, ένα σωρό κατά. Ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 6, χωρίς τη ψηφοφορία, το πρώτο μέρος πρώτα υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Το πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14 το πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. Να το ελέγξουμε. Να ελέγξουμε το δεύτερο μέρος. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Mm. Ähm, Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Αυτό με εκπλήσει. Τροπολογία 15, το πρώτο μέρος. Ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Κατόπιν έχουν με μία προφορική τροπολογία των πρασίνων. Θα ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και κατόπιν το δεύτερο μέρος. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και κατόπιν φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. 41 ψηφοί υπέρ, 5 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια στην Ιούτα Χάοκ. Χαιρόμαστε που έχουμε μαζί μας ένα τόσο σημαντικό μέλος της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστούμε πολύ. Κατόπιν φτάνουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ρίωση συν διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί του χρόνου τον Ιούνιο. Συμφωνήσαμε να κάνουμε μια προφορική ερώτηση σε συνδυασμό με ψήφισμα. 185 τροπολογίες έχουμε και 15 της Επιτροπής Ανάπτυξης. Ευχαριστώ όλους τις, ε, τους συνεισηγητές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την ε, ψηφοφορία. Οι τροπολογίες 39 και 100 ε, έχουν αποσυρθεί. Θα ξεκινήσουμε με την παράγραφο 1, τροπολογία 26. Καρτί οτάρ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε αυτό τη 30. Beendet ist Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 31, 32 και 33 που είναι όμοιες. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος. Ποιος είναι υπέρ κατά, άποχες, εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές. Να το ελέγξουμε αυτό, το δεύτερο μέρος. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Φτάνουμε στο, τέταρτο μέρος, διότι το τρίτο ήδη καλύφθηκε. Το τέταρτο μέρος ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. ένα, πρώτο μέρος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές Δεν σηκώνουν όλα τα χέρια να το ελέγξουμε. Την 44 ελέγχουμε. Ah. Λήξη της ψηφοφορίας. Ο, απορρίπτεται. Λυπάμαι. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 με προφορική τροπολογία υπέρ. Παρακαλώ. Απλά ήθελα να πω ότι είμαστε κατά της προφορικής ε, τροπολογίας, αλλά είμαστε υπέρ της αρχικής, τροπολο... της αρχικής γραπτής τροπολογίας όπως προτάθηκε. Έτσι υπάρχει αντίρρηση και γι' αυτό θα ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο χωρίς την προφορική τροπολογία, έτσι λένε οι κανόνες. Ε, ψηφίζουμε λοιπόν το αρχικό κείμενο της τροπολογίας. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύε ΕΠΤΑ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50, ε, χωριστή ψηφοφορία σε τρία μέρη. Το πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το τρίτο μέρος, υπέρ, κατά, Άποχες εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Η 5 καταπίπτει. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60 χωριστή ψηφοφορία, το πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64 και 65 είναι όμοιες υπέρ κατά Αποχές απορρίπτονται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 70 χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 71. Το πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71 το δεύτερο μέρος υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται το τρίτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 το πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Εντάξει. Να να το ελέγξουμε, την 90. Und beendet. Abgelehnt, ne? Απορρίπτεται. ΔΒ10 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 91 υπέρ κατά αποχές δεκτή 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή δεύτερο τμήμα υπέρ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 Πέρασε προφορίες. Δεκτή. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 100 έχει αποσυρθεί. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 102 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές δεκτή 102 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή 103 υπέρ κατά αποχές δεκτή 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές δεκτή 106 υπέρ κατά αποχές δεκτή Εκατόν οχτώ υπέρ κατά αποχές δεκτή 109 υπέρ κατά αποχές δεκτή 111 υπέρ κατά αποχές δεκτή 110 υπέρ κατά αποχές δεκτή 112 υπέρ για την 110 ε, θέλετε έλεγχο έλεγχος για την 110 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 113 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 115 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 117 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 119 υπέρ κατά αποχές δεκτή 121 υπέρ κατά αποχές δεκτή 120 υπέρ κατά αποχές δεκτή 122 υπέρ κατά αποχές δεκτή 124 υπέρ κατά αποχές δεκτή 123 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό 125 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 126 Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές δεκτό 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 Δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. <clears throat> Αποχές δεκτό επίσης. 1.30 μπελία υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεκτή. 1.31 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές δεκτή 134 υπέρ κατά αποχές δεκτή 135 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή 136 υπέρ κατά αποχές δεκτή 137 υπέρ κατά αποχές δεκτή 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 υπέρ κατά άποχες δεκτή 140 μπελιέ υπέρ κατά άποχες δεκτή 141 υπέρ κατά αποχές δεκτή 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται με τις υγείας σας. 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτσες. <laughs> Υπάρχει γρήπη που κυκλοφορεί εδώ. 146 υπέρ. Κατά απόχες απορρίπτεται. Δεύε 13 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. 147 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται. 148 υπέρ κατά απόχες δεκτή. tv 15 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 152 μπελία και πάλι υπέρ. Κατά. Ξέχασα δύο τροπολογίες. 150 μπελιέ πρώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 151. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απολύτω. 1,52 μπελιέ όμως. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 153. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 161 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά για μια ακόμη φορά εκ μέρους των πρασίνων. Είμαστε υπέρ της γραπτής τροπολογίας αλλά κατά της προφορικής που περιορίζει το κείμενο διότι η αξιολόγηση χρειάζεται για όλες τις τεχνολογίες, όχι μόνο για έναν ειδικό τομέα. Έχουμε αντίρρηση λοιπόν κατά της ε, προφορικής ε, τροπολογία οπότε ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο. Ποιο είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 172, 173, 174 είναι όμοιες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 183 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 185 υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 το πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ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 αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές επίσης εγκρίνεται. Έτσι φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία. λήξη της ψηφοφορίας. Χαίρομαι πάρα πολύ. 47 υπέρ, ε, καμία ψήφος κατά, καμία αποχή. Εγώ νόμιζα ότι θα βγαίναμε 50-50, αλλά ε, ακόμα καλύτερα έτσι. Ε, θερμά συγχαρητήρια στους συνεισηγητές. Υπήρχαν αντιρρήσεις όσον αφορά τις λεπτομέρειες, ε, αλλά γενικά υπήρχε συνένεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτές ήταν οι ψηφοφορίες. Έχουμε τώρα δύο σημαντικά νομοθετικά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε σήμερα το απόγευμα. Περνάμε στο σημείο 5 της ημερησίας διάταξης για την οδηγία ΒΗ δηλαδή για τα ε, ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα. Όσοι δεν θέλουν να παρακολουθήσουν, σας παρακαλώ ηρέμους και ησύχως να αποχωρήσετε. Τα πηγαδάκια εκτός αιθούσης. Εντάξει. Όσοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση, σας παρακαλώ να συνεχίσετε τις τόσο ενδιαφέρουσες ανταλλαγές απόψεων εκτός της αιθούσης. Και αυτό ισχύει ακόμα και για τους πρασίνους. Ευχαριστώ. Ο Καρλ Χάιντς Φλόρενς είναι ο εισηγητής μας για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα. Έχουμε ήδη εγκρίνει τη στρατηγική για την αποτελεσματικότητα για τα θέματα αυτά και πιστεύω και ελπίζω ότι όλα αυτά στα επόμενα χρόνια θα μπορέσει να ενσωματωθεί αυτή η λογική στην σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, όπως θα ακούσουμε και από τον εισηγητή, είχαμε κάποιες δυσκολίες με το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά την νομοθετική διαδικασία. Φαίνεται ότι έχουμε πάρα πολύ περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά δίνω στην αρχή το λόγο στον εισηγητή, μετά στους κοιόδης και μετά στους άλλους ενδιαφερομένους. Τον Καρλ Χάινς Φλόρενς λοιπόν δίνω το λόγο για να, παρακολου παρουσιάσει την κατάσταση των πραγμάτων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γιο. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους από τις πολιτικές ομάδες που συνέβαλαν σε αυτό το έργο, όπως και τους συνεργάτες μου που με βοήθησαν πάρα πολύ. Και όλα αυτά είναι απαραίτητα για τον εξή λόγο. Όλοι μας είχαμε μια κοινή ιδέα για τα θέματα αυτά σε σχέση με τα απόβλητα, με μικρές διαφοροποιήσεις. Μπορούμε να συζητήσουμε για τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρουμε όλοι ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παίζει ένα σημαντικό ρόλο, ιδίως στη χώρα μου, ο αρμόδιος επίτροπος έχει παρουσιάσει ποια ήταν η θέση που ανέλαβε το Συμβούλιο. Είχε την χαρά να συζητήσει τη στρατηγική για τους για τους πόρους με το Συμβούλιο και τόνισε πόσο σημαντική είναι αυτή η πολιτική υλικών πόρων με, ε, το Συμβούλιο. Όταν φτάσαμε στο Συμβούλιο, ε, στο σημείο 2 που ήταν τα ηλεκτρονικά θέματα, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά, υπήρξε απόλυτη έλλειψη συμφωνίας. Υπήρξε ένα χάος. Όλα αυτά τα οποία είχαμε πετύχει σε σχέση με τις πρώτες ύλες, με τους βασικούς πόρους, αυτή ουσιαστικά δεν ευδοκίμησε. Το Κοινοβούλιο πριν από 7-8 χρόνια είχε ήδη ζητήσει να ακολουθεί μια σωστή γραμμή όταν είχαμε εγκρίνει μια οδηγία για τα απόβλητα από τα αυτοκίνητα, αλλά τα πράγματα τώρα δεν είναι τόσο εύκολα. Και θα μιλήσω και στις τροπολογίες τώρα. Εμείς έχουμε απόλυτο δίκιο σε αυτή την περίπτωση γιατί έχουμε κατανοήσει ότι οι πρώτες ύλε είναι απαραίτητες και για τις επερχόμενες γενναίες και άμα θέλουμε να ελέγξουμε την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να έχουμε πραγματικά καινοτόμα συστήματα και συσκευές. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε κέρυες πρώτες ύλε για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των συσκευών μας. Επομένως η ανάκτηση των πρώτων υλών των σπανίων πρώτων υλών είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν πρέπει λοιπόν μονάχα φραστικά να αναφερόμαστε στα θέματα αυτά, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα βήματα. Αυτό μας φέρνει σε σύγκρουση με το Συμβούλιο. Θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι λοιπόν έναντι του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο σε κάποια σημεία έχει κάνει κάποιες θετικέ ενέργειες για να μην μπορούμε να πούμε ότι, τα, ότι δεν κινήθηκε καθόλου αλλά μετά από την ε, συζήτηση για την έκθεση αυτή θα πρέπει το Συμβούλιο να κινηθεί περισσότερο, να κατανοήσουν και οι μεγάλε χώρε τη Ευρώπη ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου. Όπω συζητήσαμε και μεταξύ των σκιωδών εισηγητών και εμένα, υπάρχει και το θέμα τη ε, ευθύνη των Ευρωπαίων παραγωγών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και κάτι το οποίο πρέπει να είναι σαφέ είναι το εξή, ότι εδώ και 20 χρόνια έχουμε μια εσωτερική αγορά Κάθε μικροπαραγωγός συσκευών στην δική μου περιοχή, παραδείγματος στην Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, πρέπει να εξασφαλίσει την έγκριση των ε, προϊόντων που παράγει σε 27 χώρες. Και εδώ μιλάμε για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Πρέπει να έχουμε λοιπόν το θάρρος ενώπιον του μέλλοντος να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες οι οποίες ανοίγονται μπροστά μας. Δυστυχώς το Συμβούλιο είναι εναντίον μιας κοινή ρύθμισης. Αυτό μας κοστίζει 60 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο γιατί υπάρχουν 27 διαφορετικές διαδικασίες έγκρισης αυτών των προϊόντων. Υπάρχει στη συνέχεια το θέμα της ανακύκλωσης το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί. Για μας η σφαίρα εφαρμογής αυτού του νομοθετήματος είναι πάρα πολύ σαφής. Θα πρέπει να έχουμε ένα ανοιχτό χώρο για όλα αυτά τα προϊόντα και αυτή την οδηγία, αλλά θέλουμε να υπάρξει και ανοιχτό πλαίσιο. Αυτό το ανοιχτό πλαίσιο βέβαια δεν είναι άμυρο προβλημάτων όπως και τα κλειστά πλαίσια. Ξέρουμε λοιπόν οι φίλοι μου οι πράσινοι ποια είναι τα προβλήματα Πολλές φορές ένας μεγάλος γερανός, ο οποίος σηκώνει τόνους, βασίζεται σε ένα μικρό ηλεκτρονικό ή ηλεκτρικό μοτεράκι. Επίσης, υπάρχει και το θέμα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που έχει συμπεριληφθεί σε αυτή την οδηγία. Εγώ έχω αγωνιστεί για μια θελοντική συμφωνία για τα θέματα αυτά και με έχει παρακολουθήσει μέχρι στιγμής η Επιτροπή Περιβάλλοντος και η παραγωγή των ηλιακών συλλεκτών στην ε, Ευρώπη δεν έχουν ακόμα καταφέρουν να μας πείσουν ότι μπορούν να το κάνουν αυτό με έναν τρόπο ο οποίος είναι θελοντικός χωρίς κάποια δεσμευτική ε, νομοθεσία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πραγματικά ανάληψη ευθύνης από τις επιχειρήσεις αφήνουν τα πράγματα να πηγαίνουν από μόνα τους. Δεν μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε αυτή την αντιμετώπιση που έχουν. Γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε μια διαφορετική πρόταση. Είναι γεγονός ότι θα, θα ενταχθούν τα φωτοβολτιακά πάνελ μέσα στην οδηγία αυτή. Ε? εκτός μικροφώνου σχόλιο για κομμουνιστικού χαρακτήρα διαδικασίες μεταξύ Προέδρου και Φλόρεντς. Το θέμα πάντω είναι το πώς θα μπορέσει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ανωνυμία σε σχέση με τα στοιχεία αυτά. Η Σουηδία μαζεύει 16 κιλό, κιλά αποβλήτων ανακάτοικο, η Ιταλία μόνο 4, αλλά η Κομισιόν δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί είναι τελείως ασαφές, ασαφείς οι ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη υποστήριξη της Κομισιόν για τυποποίηση και προτυποποίηση σε σχέση με την συλλογή όλων αυτών των ε, αποβλήτων. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για τη συνεργασία μας παρεμφετικά. Επίσης οι κανόνες για να μπορούμε να εξασφαλίζουμε ότι τα προϊόντα τα οποία αγοράζονται εξ αποστάσεως θα μπορούν να ανακυκλώνονται. Γιατί άμα πάρετε κάτι από ένα ε, μαγαζί είναι απλό το να το πάτε πάλι στο ίδιο μέρος. Αλλά είναι πρόβλημα αν έχετε αγοράσει κάτι από το ίντερνετ ή οτιδήποτε τέτοιο. Πρέπει επομένως να δούμε με ποιο τρόπο στο μέλλον θα έχουμε μια καλύτερη καταμέτρηση της ποσότητας αποβλήτων που παράγεται και αυτό θα πρέπει να είναι η βάση μας για να καταλάβουμε τι γίνεται. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ένα ποσοστό των ποσοτήτων που βγαίνουν στην αγορά είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να είναι ε, τα απόβλητα. Στη χώρα μου είναι αυτό πολύ εύκολο. Αλλά άμα πάτε σε άλλες χώρες όπως στην Ανατολική Ευρώπη, ο τζίρος των επιχειρήσεων για τα θέματα αυτά δεν είναι τόσο μεγάλος. Γι' αυτό εμείς έχουμε ακολουθήσει ένα διαφορετικό υπόδειγμα ότι θα πρέπει να καταμετράτε η κατανάλωση σε ηλεκτρισμό αυτών των αποβλήτων για να μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο, πόσα απόβλητα έχουμε δημιουργήσει. Υπάρχουν ήδη κάποια κράτη-μέλη όπως η Αυστρία που έχουν πλησιάσει ήδη τους στόχους μιας ανακύκλωσης ύψους 80%. Το κυριότερο έλλειμμα αυτή τη στιγμή για την οδηγία αυτή για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα είναι η παράνομη εξαγωγή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Χιλιάδες κοντέινερ φεύγουν κάθε μήνα από την Ευρώπη. Έχουμε αναπτύξει κοινού κανόνες με την Κομισιόν. Έχουμε ζητήσει να υπάρξει αντιστροφή του βάρους αποδείξεων και εδώ δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα περιθώριο για να παρακάμπτονται οι κανόνες. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει αντιστροφή του βάρους απόδειξης ώστε να αποτρέψουμε τις παράνομες εξαγωγές ε, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων δυνητικά υψηλής αξίας σε πρώτες ύλες. Και τέλος, για το θέμα της ε, χρηματοδότησης. Δεν έχω καταθέσει καθόλου τροπολογίες και ακολουθώ αυτά τα οποία θα δεχτεί η Επιτροπή μας, αλλά εάν οι συντάκτες των τροπολογιών μπορούν να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την άποψή τους, μπορούμε, μπορώ και να τους υποστηρίξω περισσότερο. Υπάρχουν τώρα ορισμένοι κλάδοι της βιομηχανίας οι οποίες βλέπουν την τάση μας να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Μα πάντα έρχεται η βιομηχανία και μας λέει αυτά που κάνετε είναι υπερβολικά γραφειοκρατικά. Θέλουν να μειώσουν στο μισό αυτά τα οποία κάνουμε, μετά έρχονται άλλοι βιομηχανικοί όμιλοι και θέλουν να μειώσουμε ακόμα περισσότερο. Παραμένει λοιπόν το ανοιχτό αυτό ερώτημα κύριε Πρόεδρε, κατά πόσο στο μέλλον τα κινητά τηλέφωνα ή τα σεσουάρ ή οι ξυριστικές μηχανές, αν όλα αυτά θα μπορεί κανείς να τα δίνει πίσω σε ένα μαγαζί, ακόμα και αν δεν αγοράζει παράλληλα ένα καινούριο προϊόν, μπορεί κανείς να έχει μια διαφορετική άποψη για τα θέματα αυτά. Και πολλοί μου λένε ότι ε, θα έρχεται ένα πελάτη στο μαγαζί μου, εγώ κάνω ό,τι μπορώ, όχι μόνο να πάρω αυτό που θα μου δώσει, αλλά να του πουλήσω κάτι. Λοιπόν, πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Ευχαριστώ πολύ, κατά τα άλλα. Ευχαριστούμε πολύ, Καρλ Χάινς Φλόρενς. Βέβαια ε, τα καταστήματα είναι καταστήματα, δεν είναι χωματερές ε, ούτε αποθήκες πρώτων υλών. Ε, θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πού είναι καλύτερο να γίνεται η συλλογή. Περνάμε στους κοιόδης εισηγητές. Τέσσερα λεπτά ο καθένας για να μπορέσουμε να παραμείνουμε εντός του χρονοδιαγράμματος. Η Κατερίν Φανμπραντ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ συμμετέχω εδώ και πολύ καιρό στην επεξεργασία αυτού του ντοσιέ. Και πιστεύω ότι θα πετύχουμε αρκετά πράγματα, αρκετές πρόοδους από ό,τι πιστεύαμε στην αρχή με αυτή την πρόταση. Βέβαια στο Συμβούλιο τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Ο εισηγητής έχει δίκιο όταν λέει ότι πρέπει να επανέλθουμε στις αρχικές ε, αξίες. Γιατί αυτή η οδηγία. Αυτή η οδηγία έχει ως στόχο τη διαχείριση των αποβλήτων. Εδώ όμως τώρα πια δεν πρόκειται μόνο για διαχείριση, αλλά και η απαραίτητη οικονομική βασικοί στόχοι διαχείρισης πρώτων υλών να αναφέρονται. Το Κοινοβούλιο πέτυχε συνένεση. Θέλουμε μια φιλόδοξη αντιμετώπιση αυτής της οδηγίας. Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα να καλύπτονται από το εφαρμοστικό πεδίο. Να γίνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανακομιδή για να πετύχουμε τους στόχους μας στον τομέα των αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Πρέπει να προσέξουμε ώστε να μπορεί με απλό τρόπο να ξεφορτώνεται ο καταναλωτής αυτά τα απόβλητα και να είναι σίγουρος ότι θα ανακυκλώνονται ας πούμε ηλεκτρικές οδοντόπουρτσες να μπορεί κανείς να τις πάει σε ένα μαγαζί και να τις αφήσει και πρέπει να επιμείνουμε όποια στάση και να έχουν τα, να κρατήσουν τα λόμπι για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Εμείς θα δούμε βέβαια τι θα γίνει, αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι μια θέση αρχής που πρέπει να συνεχίσουμε να υπογραμμίσουμε. Να υπογραμμίσουμε. Για το εφαρμοστικό πεδίο. Το ανέφερε ο εισηγητής και εγώ επιμένω. Για την ομάδα μου αποτελεί νίκη να συμπεριληφθούν στο κείμενο και τα φωτοβολταϊκά πανό για το μέλλον. Λοιπόν, αυτοί που μας ακούνε να το ξανακούσουν το μήνυμα βρίσκεστε, εντάσσεστε μέσα στο εφαρμοστικό πεδίο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί και θα πρέπει τα προϊόντα σας να τα ανακυκλώνετε και να ξαναχρησιμοποιούνται αν χρειαστεί. Και θα ολοκληρώσω ευχαριστώντας τον κύριο Φλόρεντς ε, Πάντα γίνεται αυτό από συνήθεια και βγαίνει. Αυτή τη φορά όμως τον ευχαριστώ εκ Πιστεύω ότι η έκθεσή του είναι εξαιρετική. Σεβάστηκε απόλυτα την εντολή που του ανατέθηκε, δηλαδή να κρατήσει τα κεκτημένα της πρώτης ανάγνωσης και να καταλήξει σε μια στέναρη κοινή θέση. Και κατάφερε με μπρίο, με κέφι ο εισηγητής να τα πετύχει όλα αυτά. Υποστηρίζουμε απόλυτα το κείμενό του, θα καταθέσουμε μερικές μικροτροπολογίες, πάντως ε, βρίσκεται όλη η ουσία της έκθεσης μέσα στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο Φλόρενς ασχολείται εδώ και χρόνια με ε, τα απόβλητα. Ε, Παναγιώτοφ είναι ο επόμενος και ο συζητητής. Παρακαλώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Φλόρενς και την ομάδα του για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει. Πράγματι, η πρώτη ανάγνωση ήταν μεγάλη επιτυχία με ευρία πλειοψηφία ε, που στήριξε τα πιο σημαντικά θέματα που θέλουμε να λύσουμε με την οδηγία αυτή. Χαίρομαι που σήμερα βλέπω ότι ο συνάδελφος Καρλ Χάινς Φλόρενς συνεχίζει να στηρίζει την ε, συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, στηρίζοντας τις αρχικές ιδέες του Κοινοβουλίου. Συμφωνώ με την ε, προσέγγιση για ε, εναρμονισμένη προσέγγιση της ενίας αγοράς ε, στην οδηγία αυτή. Πιστεύω ότι οι κανόνες θα πρέπει να είναι πανευρωπαϊκοί. Επιμένοντας στην ευρεία προσέγγιση και παρέχοντας επαρκή χέγγυα για την ε, καταπολέμηση της, ε, της παράνομης ε, χρήσης είναι κανόνες τους οποίους στηρίζουμε και εμείς. Γι' αυτό είναι πολύ φιλόδοξο το σύστημα επιστροφής 0 προς 1 και προσλέπω στην επιτυχία των συζητήσεων με το Συμβούλιο για να καταλήξουμε σε συμφωνία κατά τη δεύτερη ανάγνωση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε Παναγιώτοφ. Η Σαμπίνε Βίλτς. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Συμφωνώ ε, γενικά, είμαι γενικά ικανοποιημένη με την ε, πρόταση του κυρίου Φλόρενς ε, και χαίρομαι που διατηρήθηκε η γραμμή του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. Και χαίρομαι επίσης που το σχέδιο δεν προσανατολίζεται σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου στα κρίσιμα σημεία. Το Συμβούλιο λέει ότι θέλει να βελτιώσει την συλλογή των ε, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Ε, όταν όμως το διαβάζω αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τη θέση που παίρνει τώρα το Συμβούλιο. Σημειώνω από τις διαπραγματεύσεις ότι το Κοινοβούλιο με την ε, ε, ε, γενή του θέση μπόρεσε να καταλήξει σε ευρεία συνένεση. Δεν κρύβω ότι βλέπω να υπάρχουν κάποια σημεία όπου θα μπορούσε να βελτιωθεί η έκθεση του κυρίου Φλόρενς, ιδιαίτερα όσον αφορά τις εξαγωγές για παράδειγμα, αλλά γενικά είμαι ικανοποιημένη. Θα πρέπει να έχουμε ψηλές ποσοστώσεις για την ε, συλλογή. Το 85% μέχρι το 2016 είναι εφικτός στόχος. Επίσης ε, δεν ε, αναφερόμαστε στα προϊόντα βιώσιμης ανάπτυξης και επίσης ε, βλέπω να ε, σπαταλάμε τους πόρους μας ε, αυτή τη στιγμή και το Συμβούλιο δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Παντού αναφέρεται ότι οι πρώτε γίνεται γίνονται όλο και πιο ακριβέ. Πρόσφατα η Ζήμες ανακοίνωσε ότι οι οικιακές συσκευές θα γίνουν πιο ακριβές την επόμενη χρονιά διότι περιέχουν σπάνιε γέε οι οποίες ε, έχουν ε, ε, ακριβήνει μέχρι, κατά μέχρι και 3.000%. Ε, συνεχίζω να πιστεύω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε το σύστημα εθνικής καταχώρησης και στο σχέδιο που βλέπουμε μπροστά μας αναφέρεται ότι ένας εμπόρος θα πρέπει να πουλάει τα προϊόντα του σε, όλες, σε όλα τα κράτη-μέλη εφόσον έχει έδρα σε ένα κράτος μέλος. Ε, μας αρέσει η μείωση της γραφειοκρατίας, ε, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος ε, να μην μπορούν να, αποδοθούν ευθύνες στις εταιρείες αυτές εάν δεν υπάρχει κάποιος ε, σε κάθε κράτος μέλος. Εγώ πιστεύω ότι κάθε παραγωγός ε, που θέλει να πουλήσει ε, τα προϊόντα του σε μια χώρα θα πρέπει να έχει και μια έδρα εντός της χώρας αυτής. Ε, και επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε τα νανοηλικά να έχουν ξεχωριστή μεταχείριση. Η νανοτεχνολογία δεν έχει αποδείξει ακόμα ότι είναι ακίνδυνη. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη από την Γερμανία που ασχολείται με το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν και οι υπόλοιποι ομιλητέ. Σα παρακαλώ να παραμείνετε στα δύο λεπτά. Ο Ρίχαρτ Ζέμπερ είναι ο πρώτο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να συγχαρώ τον Καλ Χάιντ Φλόρεν για τα θαυμάσια εργασία που έχει φέρει σε πέρα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω πόσο σημαντικό είναι να είμαστε προσεκτικοί με τη χρήση των πρώτων υλών και να εξασφαλίσουμε την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους Πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές και να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις αδυναμίες μας στις διαδικασίες της ανακύκλωσης. Παράλληλα όμως με την οδηγία αυτή θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο για το πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την τεχνολογία μας ακριβώς για να έχουμε μια καλύτερη ε, επαναξιοποίηση των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών. Χρειαζόμαστε μια βάση η οποία, ελέγχου η οποία θα εξασφαλίσει ότι δεν γίνεται παράνομη ε, εξαγωγή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών υλικών, αλλά συγχρόνως πρέπει να βελτιώσουμε και τις τεχνολογίες μας. Υπάρχουν πολλοί φιλόδοξοι στόχοι οι οποίοι αναφέρονται, αλλά επιπλέον τα μεγάλα κράτη-μέλη θα πρέπει να, κάνουν τους πολίτες να κατανοήσουν ότι η ανακύκλωση έχει νόημα. Υπάρχει μια εκπαιδευτική διαδικασία που πρέπει να επομισθούν τα κράτη-μέλη και η ίδια η Κομισιόν ευνοώντας τις βέλτιστες πρακτικές θα πρέπει να καταδείξει <clears throat> ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση γιατί δεν έχει νόημα να έχουμε σε ορισμένε περιπτώσει πολύ ψηλό ποσοστό συλλογή και ανακύκλωση και σε άλλε περιπτώσει πολύ χαμηλό πρέπει η Κομισιόν να εξασφαλίσει, εάν θέλουμε αυτού του στόχου να του επιτύχουμε, να εξασφαλίσει ότι όλα τα κράτη-μέλη θα εφαρμόσουν με πιο ομοιόμορφο τρόπο αυτού του κανόνε. Ένα μικρό σημείο το οποίο θα ήθελα επίση να αναφέρω, Όπω τόνισε ο, ο πρόεδρός μας, τα μαγαζιά που πουλάνε ηλεκτρονικέ και ηλεκτρικέ συσκευέ, δεν έχω ματερές, θα πρέπει να υπάρχουν πραγματικά μεγάλε, ε, να υπάρχουν διαδικασίες Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε ένα κεντρικό χώρο να δίνουν τα απόβλητά τους και όχι να επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο τα καταστήματα εμπορίας. Αυτό δεν είναι δικαιολογημένο. Και επίσης αναφέρθηκε το θέμα της ευρωπαϊκής έγκρισης. Και η ευρωπαϊκή <clears throat> έγκριση είναι σημαντική, αλλά εδώ το θέμα είναι να υπάρχει δυνατότητα να παρεμβαίνει κανείς. Δεν σημαίνει δεν έχει νόημα σε κάποιες χώρες να υπάρχει μια έγκριση η οποία οδηγεί σε περαιτέρω κόστος και αλλού να μην υπάρχει κάτι τέτοιο και να υποχρεώνεται κανείς να υπόκειται σε αυτές τις διαδικασίες. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το εξηγήσουμε στους παραγωγούς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Γι' αυτό υπάρχει η, 52, η τροπολογία 52 δεν πρέπει να παραμελήσουμε το θέμα της, κοινωνικοποίη, της, κοινο, της ανακοίνωσης και της επικοινωνίας για τα θέματα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικοινωνεί η Κομισιόν με όλους τους εμπλεκόμενους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να τους εξηγεί όλα αυτά. Επίσης και οι καταναλωτές θα πρέπει να αναλάβουν κάποια ευθύνη. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει νόημα να συλλέγουμε όλα τα υλικά από το σπίτι. Θα πρέπει και ο καταναλωτής να συμβάλλει στο να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Νομίζω πάντως ο Καρλ Χάιντς Φλόρενς έχει ακολουθήσει εν γέννη τη σωστή γραμμή που υποστηρίζει το Κοινοβούλιο μας εδώ και δεκαετίες. Ευχαριστώ. Η κατάσταση είναι φυσικά διαφορετική από κράτος μέλος σε κράτος μέλος στη Γερμανία. Εάν έχουμε ένα πέραν των σκουπιδιών και ένα κάδο που βάζουμε τα ηλεκτρονικά αγαθά τα οποία έχουν ακόμα κάποια αξία όπως είναι όχι μόνο τηλεοράσεις και ε, άλλα ηλεκτρονικά υλικά αλλά και, και μπαταρίες βλέπουμε ότι με το να υπάρχει μια τέτοια εκπαίδευση του καταναλωτή οδηγεί σε μεγαλύτερο ποσοστό συλλογή. Αν πρέπει όλα να γίνονται με τα να πηγαίνει τα απόβλητα στο κατάστημα, μειώνεται αυτό το αυτή η υπευθυνοποίηση και το γεγονός ότι συμβάλλει. Θα πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε για να έχουμε ενιαίες ποσοστώσεις ότι η βιομηχανία είναι πράγματι σε θέση να κάνει μια επιλογή <clears throat> και διαλογή των υλικών. Η Κορίν Λεπάζου. Και εγώ κύριε Πρόεδρε θα συγχαρώ τον εισηγητή. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο και πολύ καλό κείμενο και χαίρομαι που ε, συμπεριέλαβε τη συναντήληψη Χαίρομαι που αναφέρεται και η πρόταση για τη χρηματοδότηση έγινε δεκτή από τον εισηγητή μας. Δύο μικρά σημεία. Τα μέτρα ελέγχου των εξαγωγών που θεωρώ ότι παραμένουν αδύναμα και το γεγονός ότι οι νομικές υποχρεώσεις δεν επεκτείνονται πέραν του κατόχου. Υπάρχει ένα πρόβλημα διαφωνίας όμως με το Συμβούλιο ε, του παραγωγού, συγγνώμη. Ε, υπάρχει ένα πρόβλημα όμως στο Συμβούλιο για τον πώς καθορίζουμε εμείς τον παραγωγό. Πέρα όμως από αυτά τα δύο μικροσημεία δεν έχω άλλο πρόβλημα και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς με το κείμενο. Ο κύριος Σλούτερ. Χάινς, ε, δεν χρειάζεται να γίνεις κομμουνιστής. Αν ε, συνεχίσεις όμως να γράφεις ε, τέτοιες εκθέσεις, σίγουρα είσαι πρόσδεκτος στους πρασίνους. Είμαστε ικανοποιημένοι με τη δουλειά σου. Νομίζουμε ότι σεβάστηκε απόλυτα την πρώτη ανάγνωση και έχει ε, συμπεριλάβει ε, το ανοιχτό πεδίο εφαρμογή ε, για να μπορούν να χωρέσουν και άλλα πράγματα όπως είναι το κριτήριο του 5% κλπ. Έχει ξαναθέσει όλα τα θέματα, το οποίο είναι θετικό. Ε, κάποιος είπε και νομίζω ότι ε, έχετε δίκιο ότι θα πρέπει να είναι ε, εύκολη η ζωή των καταναλωτών αλλά από την άλλη δεν θέλουμε να χάσουμε τις δυνατότητες των λιανοπολιτών να μπορούν να πάρουν πίσω τουλάχιστον τις μικρές συσκευές διότι Μπορεί να, μπορεί να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να επισκευάσει, να, να, να, επισκευαστεί το, η συσκευή του και να την πάει στο κατάστημα. Ε, αλλιώς θα πρέπει να την ξαναπάρει πίσω και να την ε, πετάξει στα απόβλητα. Αλλά ε, ίσως είναι πιο χρήσιμο να μπορεί να την αφήσει στο κατάστημα όπου την πήγε. Ε, αλλά, υπάρχει εξαίρεση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ε, ε, ένα πράγμα που θα ήθελα να φέρω είναι τα νανοηλικά. Υιοθετήσαμε μια πολύ ε, μετριοπαθή ε, τροπολογία για τα νανοηλικά. Κομισιόν περιμένω ακόμα απάντηση για την έκθεσή μου του 2009. Είμαι ακόμα γενικός, αλλά αν αργήσετε πολύ ακόμα θα, θα χάσω την υπομονή μου. Πάντως ε, είπατε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση των κινδύνων από τα νανοηλικά και όταν θα υπάρχει αυτό να συμπεριληφθεί στο παράρτημα 7. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον κανονισμό. Και τέλο. Νομίζω ότι είναι λίγο περίεργο που μιλάμε για απόβλητα. Ε, εγώ θα μιλούσα για αστικά ορυχτά, urban mining που λέμε στα αγγλικά, διότι ε, υπάρχουν πολύτιμα ορυκτά ε, σε όλα τα ε, ε, απόβλητα αυτά. Πρόκειται για πόρο, δεν πρόκειται για απόβλητα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ο Καλχάινς Φλόρενς μπορεί να προσχωρήσει τους κομμουνιστές αν θέλει είτε στους οικολόγους. Ο Πίτερ Λίζα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τα όσα είπε ο Καλχάινς Φλόρενς καθώς και ε, με τους συναδέλφους ε, που τον στήριξαν. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ περίεργη η κατάσταση. Ε, για παράδειγμα, είναι πολύ σπάνιες, οι σπάνιες Ε, Έχουμε δει ραγδαία αύξηση των τιμών και δεν είναι απλή η ανακύκλωση. Το είδα στην εκλογική μου περιφέρεια ότι βρίσκεται ακόμα σε, σε, σε, σε πολύ πρώιμο στάδιο η ανακύκλωση. Εάν ε, ε, ε, εγκαταλείψουμε όμως την ιδέα της ανάκτησης των υλικών θα κάνουμε μεγάλο λάθος. Εγώ έχω ασχοληθεί με τον φωτισμό, με τους λόγους κτλ. Και πράγματι γίνεται προσπάθεια ανάκτησης των σπάνιων γεών από τους παλιούς γλώβους. Αλλά θα πρέπει τότε να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα συλλογής. Θα πρέπει λοιπόν αυτό που ουσιαστικά γίνεται στην Ευρώπη να εφαρμοστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης θα ήθελα να συμφωνήσω με την τροπολογία 53 που έχει να κάνει με τις μικρές ε, συσκευές. Ε, την ε, είχα υποβάλει αρχικά μαζί με τον συνάδελφο Σκυλακάκη. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε σχετικό συμβιβασμό για ε, μια σειρά μικρών συσκευών ε, σε κάποιους δήμους ε, υπάρχουν κάδοι συλλογής αλλά θα πρέπει να είναι φιλική προς τον καταναλωτή και όσον αφορά τους γλώπους, τις λάμπες, τις οικονομικές, τους οικονομικούς λόπους αυτούς δεν μπορούν να τους ρίξει κανείς απλά στον κάδο θα πρέπει εδώ να γίνεται επιστροφή στο κατάστημα. Κάποιοι το κάνουν αυτό εθελοντικά και θα πρέπει να τους ε, ενθαρρύνουμε και αυτούς ε, που αντιστέκονται να τους ε, κινητοποιήσουμε περισσότερο. Θα μπορούσαμε να θέσουμε μια προθεσμία. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να λειτουργεί το σύστημα αυτό. Μία ερώτηση έχω προς τον εισηγητή που έχει να κάνει με το θέμα του φωτιστικού υλικού με την τεχνολογία LED. Ε, βλέπουμε συγχώνευση ε, των διαφόρων τεχνολογιών. Μήπως θα ήταν τότε χρήσιμο να ε, έχουμε μία κατηγορία εδώ, διότι αλλιώς θα είναι δύσκολο να χειριστούμε το σύστημα εάν έχουμε κάποια προϊόντα όπου υπάρχει συγχώνευση των διαφόρων τεχνολογιών. Σύμφωνα με τα σχέδιά μας, πρόκειται για χωριστές κατηγορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η Σοφία Κονή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ παίρνω το λόγο για μένα και εκπροσωπώντας την Φρανσουάς ε, Γκροστέτ που δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα. Συγχαίρω τον κύριο Φλόρεντς για την ποιότητα της έκθεσης του που είναι πολύ φιλόδοξη. Πρόκειται για μια ουσιαστικότατη έκθεση από τα 9 εκατομμύρια τόνων αποβλήτων ε, ελάχιστα σήμερα συλλέγονται σωστά. Για τις διασυνοριακές μεταφορές ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων πρέπει να προβλέψουμε κάτι και θα πρέπει η παραγωγή να και οι ε, πολιτές, οι διανομής να ε, ορίσουν ένα σύστημα ανακομιδής αυτών των ε, αποβλήτων. Θα πρέπει επίσης ε, να θέσουμε και θέματα προσωπικής διαπαιδαγώγησης στην ανακύκλωση, με τα πορητά τηλέφωνα, πόσοι δεν κρατάμε ε, παλιά φορητά τηλέφωνα και δεν τα ανακυκλώνουμε. Άλλα σημεία όπως είπε η Κορίν Λεπάζο, ο ευρωπαϊκός ορισμός του παραγωγού. Εάν θέλουμε εμείς διοικητική απλούστευση για αυτό το θέμα και να εναρμόσουμε τα εθνικά μητρώα παραγωγών, αυτός ο ευρωπαϊκός ορισμός για τον παραγωγό μας φαίνεται επικίνδυνος. Η Φρανσουάς Γκροστέτ το θύμισε κατά την πρώτη ανάγνωση. Ένα λοιπόν έχουμε τον Ευρωπαίο παραγωγό που υπόκειται στην ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και των αποβλήτων διότι τότε το απόβλητο μπορεί κάλλιστα να κυκλοφορεί με περιβαλλοντικούς κινδύνους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυσκολίες επίσης Ε, οπότε ε, μπορεί να δημιουργηθούν και προβλήματα ε, ρήπανσης πρέπει δεν υπάρχει μετά άνοιχνες, άνοιχνευσιμότητα όταν έχουν τα πόβλητα περάσει σε έναν τρίτο και επίσης δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε ό,τι να είναι από την οδηγία. Το θέμα της ανακύκλωσης, ποσοστό ανακύκλωσης αξιολόγησης αλλά να είναι στόχοι εφικτοί. Η διαφάνεια του κόστους ανακύκλωσης και ανακομιδής, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε, αντίθετα από αυτό που είπε ο κ. Σλίτερ, να σκεφτούμε τι κάνουν οι μικροί λιανοπολιτές και οι μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν τα μέσα ούτε τον ε, χώρο για να μας διασφαλίσουν με αυτή την ανακομιδή και για την κατηγορία τώρα του ηλεκτρονικού ε, και ηλεκτρικού εξοπλισμού γιατί να ξεχωρίζουμε τα φωτιστικά από τις λάμπες πολλές φορές και με την τεχνολογική πρόοδο είναι το ίδιο πράγμα. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε και μια άλλη φορά με τον συνάδελφο Φλόρεντς. Η Καρίν Κάλεμπαχ. Μετά από όλα αυτά από αυτούς τους ε, ένους είναι σαν να μην έχει να αλλάξει τίποτα ο κύριος Φλόρενς. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε κάποια δυνατότητα να λειτουργήσουν οι μικρές επιχειρήσεις. Εγώ έρχομαι από το μάρκετινγκ καταρχήν και ξέρω πόσα εκατομμύρια δίνονται για αυτή την πρώτη επαφή με τον καταναλωτή, με τον αγοραστή. Πρέπει λοιπόν να είναι σαφές ότι μιλάμε για μικρές συσκευές, να μην πηγαίνει κανείς με μια ολοκληρή τηλεόραση και να την πετάει σε ένα κατάστημα. Εγώ έχω μια μικρή ε, αίτηση, εγώ έχω μια δυσκολία με την έκφραση των ε, αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν σε αυτή την ε, οδηγία. Αυτό πώς θα μπορούσαμε να το καθορίσουμε λιγάκι καλύτερα. Ε, ο κ. Καμπράντη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι ο μόνος που δεν πήρε το λόγο, γι' αυτό είπα να τον πάρω. Και να μιλήσω για να επενέσω κι εγώ τον κύριο Φλόρεντς όχι μόνο για την ποιότητα αλλά και για την ταχύτητα διότι θέλει να προχωρήσει γρήγορα αυτή την οδηγία δεν πρέπει να ξεπεραστούμε από την πράξη, από την πρακτική εγώ κάθε μέρα ασχολούμαι με θέματα πρώτων υλών και σε μερικά χρόνια θα έχουμε έναν μικροεπιχειρηματία ο οποίο θα στήσει την επιχείρηση του για να μπορεί να και όλοι θα τον πληρώνουν για να μαζεύει αυτά τα απόβλητα. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα για να βρούμε γρήγορα συμφωνία με το Συμβούλιο. Εκπλήσωμε με τον τρόπο που δρά το Συμβούλιο. Ο στόχος για την αποτελεσματικότητα των κονδυλίων είναι πολύ σημαντικό σύμφωνοι. Όταν πρόκειται όμως για συγκεκριμένα μέτρα δεν κάνει τίποτα. Στη συνέχεια κύριε Πρόεδρε, αυτοί που παραπονιούνται για το κόστος και τα ρίσκα της ανακομιδής αλλά και αυτά τα εγώ τα έχω στο τραπέζι μου. Πάντοτε οι ίδιοι είναι αυτοί οι οποίοι τελικά μαζεύουν τα απόβλητα. Πρέπει να τα πούμε διαφορετικά όλα αυτά, να τα δούμε κάπως διαφορετικά, διότι όλα τα στοιχεία που βρίσκονται μέσα στα μηχανήματα αυτά είναι πολύτιμα και δεν μπορούμε να τα συλλέξουμε όλα. Η Κομισιόν τώρα έχει το λόγο. Πέντε λεπτά αν μπορείτε για βέλτιστη χρήση του χρόνου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον εισηγητή για την έντονη εργασία που το έχει φέρει σε πέρας. Ξέρουμε όλοι μας ότι αυτή η οδηγία είναι ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο μας για να έχουμε μια Ευρώπη με μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη χρήση των φυσικών πόρων και αυτό αντανακλάται στην ε, έντονη προσπάθεια που καταβάλουν τα τρία θεσμικά όργανα. Σε την πρώτη ανάγνωση κάθε θεσμικό ε, όργανο έχει μία ισχυρή, μια στεναρή θέση, αλλά χωρίς κοινή συμφωνία. Πηγαίνοντα τώρα στη δεύτερη ανάγνωση, όλα τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να προβούν σε κάποιες παραχωρήσεις και υποχωρήσεις είναι αυτό το έργο ενώπιόν μας, αλλά είμαι πεπισμένοι ότι θα φτάσουμε σε μια συμφωνία που θα υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει πιο αποτελεσματική <clears throat> κοινωνία στη χρήση των φυσικών πόρων. Θα ήθελα να αντιδράσω τώρα κύριε Πρόεδρε σε μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο έκθεση και κάποια από τα οποία ανέφερε ο κύριο Φλόρεν. Ο εισηγητή προτείνει καταρχήν η Επιτροπή Περιβάλλοντος να υποστηρίξει τη συμπερίληψη των φωτοβολταϊκών πάνελ στο, στην εμβέλεια της οδηγίας. Η Κομισιόν μπορεί να δεχτεί ότι η συλλογή και η επεξεργασία των φωτοβολταϊκών πάνελ θα πρέπει να εξασφαλιστεί. Μετά την τελευταία ψηφοφορία στην ε, Ολομέλεια και την, μετά από αυτήν και μέχρι την έκθεση αυτή, η Κομισιόν έχει κάνει μια μελέτη αντικτύπου για το τι θα συνέβαινε αν συμπεριλαμβανόταν και τα φωτοβολταϊκά και η μελέτη αυτή δείχνει ότι είναι σημαντικά τα ωφέλη που θα προσποριστούμε από την ανακύκλωση και αυτών των υλικών. Το σχέδιο έκθεσης επίσης τονίζει τη σημασία να επιτευχθούν φιλόδοξοι στόχοι συλλογή σε ένα εύλογο και ορατό χρονικό οριζόντα. Και σε αυτό συμφωνεί η Κομισιόν και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες για το πώς θα πρέπει να καθοριστούν αυτοί οι στόχοι, ώστε να είναι συγχρόνως αμπίση, να είναι φιλόδοξη, ισοδίκαιη και επιτεύξιμη. Αναφέρθηκε επίση ο κ. Φλόρενς για τις παράνομες εξαγωγές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, αποβλήτων δηλαδή. Ένας από τους σημαντικούς στόχου της πρόταση τη Κομισιόν είναι να μειωθεί αυτή η παράνομη εξαγωγή ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων με το να τεθεί το βάρο αποδείξεως σε αυτού οι οποίοι προβαίνουν στις εξαγωγές. <clears throat> Ο στόχος μας είναι να υπάρξει περισσότερο φως σε μια προβληματική περιοχή, δηλαδή το πώς να εξασφαλιστεί η εξαγωγή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, αλλά να απαγορευτεί συγχρόνως η εξαγωγή αποβλήτων που καμουφλέονται πολλές φορές ως συσκευές από δεύτερο χέρι. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους θα έχουμε ένα αποδεκτό τρόπο να επιτύχουμε αυτό το σημαντικό στόχο. Η έκθεση επίσης τονίζει τη σημασία του να υπάρχει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών ώστε η οδηγία να μην οδηγήσει σε διοικητικό άγχος το οποίο θα επηρεάσει την κοινή αγορά για, τα ηλεκτρικά και, για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Και πάλι είναι μια προσέγγιση την οποία τη την ε, αποδέχεται απόλυτα η Κομισιόν. Και αυτό αφορά παραδείγματος χάρη την περίπτωση διαμεθοριακών εξαποστάσεως πωλήσεων. Η υποχρέωση του διανομέα να πάρει πίσω τα υλικά αυτά, τις ηλεκτρονικέ αυτέ συσκευέ, αυτή είναι η πρόταση του εισηγητή. Η Κομισιόν δεν έχει αντίρρηση με μια τέτοια πρόταση. Η Κομισιόν, σύμφωνα με τον εισηγητή, λέει ότι πρέπει να δώσει στις υπηρεσίες τυποποίησης την ε, εντολή να δημιουργήσουν πρότυπα για τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρονικά απόβλητα. Εμείς ήδη μέσα στο πρόγραμμα Live προσπαθούμε να προχωρήσουμε στην ε, δημιουργία τέτοιων προτύπων και έχουμε έρθει σε επαφή με αυτό το φορέα. Κάτι ακόμα που θέλω να υπενθυμίσω εν συντομία είναι ότι οι συζητήσεις για αυτή την οδηγία γίνονται βάσει της ε, συμπεφωνημένης συμφωνίες για την αναδιατύπωση μιας οδηγίας. Αυτό δεν επιτρέπει να υπάρξουν αλλαγές στο, σε θέματα που δεν είχαν αναφερθεί στην αρχική πρόταση της Κομισιόν. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος τόνισε στην ε, συζήτησή της την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε και την επίπτωση σε οικονομικό επίπεδο για τους κατασκευαστές τέτοιων προϊόντων. Και το επαναλαμβάνει η εκθέση του κ. Φλόρενς, αλλά θέλω να τονίσω ότι παρά το γεγονός ότι συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι αυτό είναι μια σημαντική ιδέα, δεν περιλαμβανόταν στο πλαίσιο τη αναδιατύπωση τη οδηγία. Κάτι άλλο που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Κομισιόν είναι ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο πλαίσιο, στο σφαίρα εφαρμογή τη ε, της οδηγίας θα πρέπει να γίνει μόνο μετά από μια εξέταση, μια μελέτη αντικτύπου. Θεωρούμε ότι όλε οι αποφάσει μα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικέ γνώσει και πραγματικά στοιχεία. Αυτή πρέπει να είναι η βάση μας λοιπόν και να κάνουμε μια συζήτηση για την αλλαγή στην εμβέλεια αυτή τη οδηγία μόνο όταν έχουμε μια έκθεση αντικτύπου για τα θέματα αυτά. Για να πέρα τόσο κύριε Πρόεδρε, όπω είπα και στην αρχή, έχουμε πολλά πράγματα να πράξουμε, αλλά είμαι πεπισμένη ότι μπορούμε από κοινού να επιτύχουμε στο εγχείρημα αυτό και μπορείτε να βασιστείτε στην Κομισιόν να σας υποστηρίξει και να διευκολύνει αυτό το εγχείρημα όταν είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκούλοφ. Για τις εξηγήσεις που δώσατε εξ ονόματο της Κομισιόν, το Συμβούλιο τώρα μπορεί να λάβει το λόγο. Κύριε Βυσνεύσκη, από την Πολωνική Προεδρία μπορεί να μας δώσει κάποια στοιχεία. Έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που έχω τη δυνατότητα σήμερα να σας μιλήσω. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα όλη τη συζήτηση. Θα ήθελα μόνο να πω ότι η Πολωνική Προεδρία θα συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη δεύτερη ανάγνωση και ελπίζουμε ότι η συνεργασία αυτή και με όλους τους άλλους ευρωπαϊκούς φορείς ε, θα διεξαχθεί ομαλά. Θα συνεργαστούμε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να τονίσω ότι η δεύτερη ανάγνωση αυτής της οδηγίας ε, ανήκει στις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία κατά τη δεύτερη ανάγνωση. Εδώ και δύο χρόνια προχωρούν οι εργασίες για το σχέδιο οδηγίας αυτό και το Συμβούλιο θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε επιτέλους να τεθεί σε ισχύ. Το σχέδιο οδηγίας αυτό συνδέεται στενά με την στρατηγική Ευρώπη 2020 και με την ενεργειακή απόδοση. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε έναν οδικό χάρτη για το θέμα αυτό, δηλαδή για την σωστή χρήση των πόρων. Η οδηγία αυτή ταιριάζει πολύ καλά στο γενικότερο αυτό πλαίσιο. και ελπίζω ότι θα αποτελέσει ένα από τα πρώτα παραδείγματα της ε, εφαρμογής της αρχής της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων. Η Πολωνική Προεδρία αγωνίζεται ώστε η οικολογική νομοθεσία πράγματι να προστατεύει το περιβάλλον και η η οικονομική διαχείριση να γίνεται με τον όσο γίνεται πιο σωστό τρόπο. Δηλαδή μα ενδιαφέρει από τη μία η πρόληψη, από την άλλη η αντιμετώπιση των αθέμητων πρακτικών. Θέλουμε να αποφύγουμε να υπάρχουν παράθυρα, να υπάρχουν γκρίζε ζώνες. Όταν ε, μιλάμε για τη συγκεκριμένη οδηγία, μιλάμε για την ε, αποφυγή παράνομων ε, τόπων διάθεσης και την παράνομη εξαγωγή των αποβλήτων. Πολύ σημαντικό είναι να διασφαλίζεται η νομική βεβαιότητα και να επιδιώξουμε απλοποίηση της νομοθεσίας ώστε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και θα ήθελα να αναφέρω ένα από τα πιο βασικά στοιχεία της οδηγίας αυτής, ε, το ανέφεραν και οι προλαλήσαντες. Πρόκειται για τον ορισμό του παραγωγού. Προτείνεται να υπάρχει ένας πανευρωπαϊκός ορισμός, ένας ορισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα κατά την εφαρμογή της οδηγίας. Έχουμε συζητήσει πολύ καιρό σχετικά με την δυνατότητα διατύπωσης ενός τέτοιου ορισμού ώστε να έχουμε ταυτόχρονα τον ευρωπαϊκό ορισμό αλλά να υπάρχει και περιθώριο για τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη όμως αντιστέκονται Ένας εθνικός ορισμός ε, του παραγωγού ε, πιστεύουμε ότι ε, επιτρέπει την καταπολέμηση της παρανομίας των παράνομων εξαγωγών, για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για τα κράτη-μέλη και πιστεύουμε ότι πρέπει να το διατηρήσουμε. Είναι σημαντικό στοιχείο αυτό για ε, την Πολωνική Προεδρία, δηλαδή να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει δυνατότητα για εθνικούς ορισμούς ε, του παραγωγού. Αυτό το πιστεύουν και άλλα μέλη του Συμβουλίου. Πάντως, όπως είπα, προσβλέπω στην καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε στενά μαζί σα. Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή. Ε, ετοιμάσατε την έκθεση αυτή ε, σε πολύ λίγο χρόνο. Στο δεύτερο εξάμεινο του χρόνου δεν έχουμε πολύ χρόνο ενώ απαιτείται χρόνος για τη συζήτηση όλων αυτών των τεχνικών λεπτομεριών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σέσκα. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι αυτό είναι μια προτεραιότητα της Πολωνικής Προεδρίας. Ξέρω ότι είναι <clears throat> επιστήμον και μηχανικός και ο αρμόδιος υπουργός θα ήθελε πράγματι να αποκομίσει κάποιο αποτέλεσμα σε σχέση με την οδηγία αυτή στο πολωνικό εξάμεινο και δίνω και πάλι το λόγο στον εισηγητή τον ευχαριστώ συλλογικά. Εφόσον όλοι σας, ευχαριστούν, απευθύνω και εγώ ευχαριστήσεις σας, Καλ Χάινς. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω σε όλα, όλα τα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν. Θα σταθώ σε μερικά ε, θέματα τα οποία νομίζω ότι είναι σημαντικά. Ο Γκαμπραντία. Εμείς έχουμε εδώ ένα μεγάλο λάθος, έχουμε κάνει ένα μεγάλο λάθος στην ε, νομοθεσία. Άμα δούμε πόση αξία καταστρέφεται στην Ευρώπη και πόση λίγη ανακυκλώνεται από τα απόβλητα, θα πρέπει να αναρωτηθούμε, φταίει η βιομηχανία ή φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις χωματερές θα πρέπει να τα επανεξετάσουμε. Αν θέλουμε να έχουμε υψηλούς στόχους ανακύκλωσης, έχει η βιομηχανία και κίνητρο να αναπτύξει τεχνολογίες και να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Εμείς όμως δεν έχουμε, δεν έχουμε αναπτύξει τέτοιους στόχους και επομένως η βιομηχανία δεν έχει ενδιαφερθεί για τα θέματα αυτά. Εμείς <clears throat> πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε και την νομοθεσία για τα θέματα αυτά. Αλλά είναι γεγονός ότι πάρα πολλά <clears throat> από αυτά τα υλικά δεν περνάνε από μία ανακύκλωση. <clears throat> Επομένως το ερώτημα αυτό το οποίο θέτεται είναι πολύ σημαντικό και το επόμενο το θέμα της συνειδητοποίησης. Πώς οι άνθρωποι αμερίμνος πετάνε στα σκουπίδια τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά αυτά προϊόντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν πολλά νέα κράτη-μέλη. Μετά από την πρώτη μεγάλη διεύνηση, μετά το 2004, που είναι πολύ καλύτεροι από τους άλλους. Είναι πολύ καλύτεροι μαθητές από τους άλλους. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, είναι και θέμα δημιουργία κινήτρων. την, ποια είναι τώρα η διαδικασία για τα προϊόντα αυτά στην Αυστρία. Από την Αυστρία είδαμε την απόδειξη ότι μπορεί να υπάρχει πραγματικά ένας φιλόδοξος αλλά και ρεαλιστικός στόχος σε σχέση με την ανάκτηση προϊόντων. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο στα νέα κρατημέλη από ό,τι στην Αυστρία, το ξέρουν όλοι. Αλλά είναι δίκαιο πιστεύω να το έχουμε αυτό ε, υπόψη μας για το μέλλον. Γιατί στα νέα κρατημέλη αγοράζονται πολλά νέα προϊόντα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουν πολλά παλιά τα οποία θα τα θέσουν σε ανακύκλωση. Για την κυρία Λεπάζ, εγώ σας προσκαλώ. Είπατε ότι έχετε ακόμα κάποιες ε, νομικές αμφιβολίες. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ. Δεν είμαι νομομαθής βέβαια, αλλά αν υπάρχουν κάποια παραθυράκια και κάποιες ελλείψεις θα ήταν χρήσιμο να μα τα, υποδο... να, τα υποδείξετε. Υπήρξαν καλές ε, ερωτήσεις ποικίλου χαρακτήρα ε, οι οποίες τέθηκαν. Εδώ θέλω στην Κομισιόν να ζητήσω να αντιμετωπίσει και το θέμα της ε, τυποποίησης. Είναι όλα ασαφή δεν υπάρχει μια σταθερή γραμμή σε σχέση με την τυποποίηση στα διάφορα νομοθετήματα που αντιμετωπίζουν εδώ πέρα. Ίσως η Κομισιόν μπορεί να είναι λίγο πιο ε, φιλόδοξη στα θέματα αυτά και εγώ θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στη δική μου χώρα που αντιστέκεται στη δημιουργία ε, ευρωπαϊκών κανόνων και ε, σε ό,τι αφορά τα ποσοστά ανάκτησης. Κοιτάξτε, εγώ έχω έρθει στο κοινοβούλιο εδώ πέρα με το όραμα μιας ε, γιγάντιας οικονομικής αγοράς και των πυλώνων που πρέπει να υποστηρίξουν την Ένωση της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν κάθε φορά που χαλάει η τηλεόρασή μας η Ευρώπη να είναι να αστοχεί και να μην έχουμε κανένα τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα το οποίο είναι ένα πολύ απλό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε κλείσει λοιπόν αυτή τη συζήτηση. 12 Σεπτεμβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. 14 4 Οκτωβρίου συγγνώμη, στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε για το θέμα αυτό, την έκθεση αυτή. Ευχαριστούμε. Ερχόμαστε στο τελευταίο σημείο της ημέρησιας διάταξης. Είναι πέντε η ώρα βέβαια και έχουν κάπως αραιωθεί οι τάξεις των βουλευτών. Παρ' όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα των βιοκτώνων. Η Κρίστα Κλάς είναι η συγγήτριά μας για το θέμα αυτό. Κυρία η συγγήτρια, και εσείς έχετε εργαστεί σκληρά για το θέμα αυτό ένα θέμα το οποίο διατρέχει πάρα πολλά προβλήματα και το αντιμετωπίζουν σε καθημερινό επίπεδο τα νοικοκυριά και οι πολίτες. Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν των πραγμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Και παίρνω στα σοβαρά αυτό που είπε ο συντονιστή μου ότι οι σημαντικοί έχουν παραμείνει στην αίθουσα. Είναι πολύ ιδιαίτερο το θέμα αυτό και όπως και η έκθεση του Κάρθενς Φλόρενς ε, έχει να κάνει με ένα θέμα για το οποίο δεν υπάρχουν ακόμα ε, ευρωπαϊκοί κανόνες. Ε, μας ενδιαφέρει η αηφόρος ανάπτυξη και γι' αυτό θα πρέπει να ρυθμίσουμε και τη χρήση των βιοκτώνων στην Ευρώπη και την σχετική αγορά. Έχουμε συγκεντρωθεί εδώ διάφοροι ειδικοί. Να ευχαριστήσω τους συναδέρφους και τη γραμματεία που έχουν συνεργαστεί πολύ καλά και κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Ε, επειδή τρέχει ο χρόνος όμως ε, πρέπει να το συστήσουμε σήμερα ε, το θέμα και ελπίζω αυτοί που δεν είναι παρόντες να διαβάσουν ή να έχουν διαβάσει την εκθεσή αυτή. Περίπου οι μισές τροπολογίες μας από την πρώτη ανάγνωση υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο και μπορέσαμε έτσι να περάσουμε κάποια από τα αιτήματά μας ε, αναφέρομαι στην αρχή της προφύλαξης, ε, την ε, σχέση με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Επίσης, τα προϊόντα υποκατάστασης για και έχουμε προθεσμία 7 αντί για 10 χρόνια. Αναφερόμαστε και στα PBT που είναι ένα κριτήριο υποκατάστασης. Δεν Υπάρχει Γίνεται ξεχωριστή αξιολόγηση κινδύνου για τα νανοηλικά, κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και έχουμε ε, συμπεριλάβει και τον ορισμό των ε, ευαίσθητων ε, ομάδων και γίνεται και διάκριση ανάμεσα στις ελαφρές τροποποίησεις και τις σημαντικές. Είμαστε λοιπόν ικανοποιημένοι με την κοινή θέση. Ε, στα ε, σημεία αυτά. Σε άλλα σημεία το Συμβούλιο έχει κάνει σημαντικό βήμα, ε, έχει μετακινηθεί σημαντικά προς τη θέση του Κοινοβουλίου. Μιλάμε για τις οικογένειες προϊόντων. Δεν, μας, δεν θα τσακωθούμε για τον όρο εφόσον εννοούμε το ίδιο με το Συμβούλιο. Έχουμε έχουν υποβληθεί πολλές ε, τροπολογίες, ε, πολλές ειδικά για μια δεύτερη ανάγνωση. Ε, αλλά αυτές οφείλονται στο ότι η κοινή θέση περιέχει αρκετές αντιφάσεις που μάλλον μπήκαν στο κείμενο λόγω της πίεσης του χρόνου. Πολλές λοιπόν από τις τροπολογίες μου είναι τεχνικής φύσης και έχουν στόχο ε, να διασφαλίσουν την συνοχή του, ε, και εντό του κειμένου και με άλλα νομοθετήματα. Και ελπίζουμε να ακολουθήσει και σχετική ε, διευκρίνηση. Όπως έχω συμπεριλάβει και εγώ τη σχετική διευκρίνηση στο κείμενό μου ότι πρόκειται καθαρά για τεχνικές τροποποίησεις. Ε, Όσον αφορά τι εφαρμοστικέ διατάξεις ε, και τις πράξεις κατεξουσιοδότηση, ήταν πολύ σημαντικό για μένα να εκφράσω τη θέση του Κοινοβουλίου. Το Συμβούλιο έχει αλλάξει πολλές από τις εφαρμοστικές διατάξεις και έτσι περιορίζει την ε, αρμοδιότητα του ε, Κοινοβουλίου. Αυτό ιδιαίτερα στο άρθρο 8α κατά την αδειοδότηση και εκεί όπου μιλάμε για τα τέλη Ε, ενώ εμεί θέλουμε με πράξη κατουσιοδότηση να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο. Η, στην κοινή θέση θετικό είναι ότι για τα βιοκτώνα που θα εγκρίνονται με απλοποιημένη διαδικασία αυτές ε, οι ουσίες θα συμπεριλαμβάνονται στο παράτιμο 1. Ε, δεν καταλαβαίνουμε όμως ότι ε, το Συμβούλιο ε, έχει κατάλογο με δραστικές ουσίες οι οποίες όμως δεν πληρούν τα κριτήρια και πέρα από αυτό όχι μόνο οι δραστικές ουσίες αναφέρονται σε παρατήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις. Εγώ πιστεύω ότι όλες οι δραστικές ουσίες με πράξεις κατοξιοδότηση και με συμμετοχή του Κοινοβουλίου θα πρέπει και που λαμβάνουν άδεια θα πρέπει να αναφέρονται ε, στον ε, κανονισμό. Ε, θα πρέπει λοιπόν να ξαναξετάξουμε τον κατάλογο των δραστικών ουσιών. Στην πρώτη ανάγνωση συμφωνήσαμε από το 2017 να υπάρχει ευρωπαϊκή αδειοδότηση όλων των βιοκτώνων με εξαίρεση αυτών που εμπίπτουν στα κριτήρια αποκλεισμού. Ε, αυτή τη στιγμή ε, το μεγαλύτερο μέρος ε, της διαδικασίας αδειοδότησης αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών και η Κομισιόν έχει πιο πολύ ρόλο συντονισμού. Η κοινή θέση προβλέπει η ενωσιακή αδειοδότηση και το πρώτο βήμα της ενωσιακής αδειοδότησης θα είναι πιο πολύ θεωρητικής φύσης διότι ήδη γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο προτείνει οικογένειες προϊόντων οι οποίες ε, δεν θα υπόκεινται σε αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης. Πέρα από αυτό, ε, το Συμβούλιο ε, εξαιρεί κάποιες, κάποια προϊόντα από τη διαδικασία αδειοδότησης. Πιστεύω από την Ευρωπαϊκή Διαδικασία Διοδότησης και πιστεύω ότι η θέση του Κοινοβουλίου αυτή είναι λάθος, διότι στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ε, καλύτερα και πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και γι' αυτό προτείνουμε τα βιοκτώνα ε, με δραστικές ουσίες που να αποκλείονται από τη διαδικασία διοδότησης ε, να μην χρειάζονται ευρωπαϊκή αδειοδότηση. Παρ' όλα αυτά προτείνω την προσέγγιση σε δύο στάδια που αφορούν τα προϊόντα τα οποία ήδη ε, έχουν ε, υποβληθεί στην ε, εξέταση προς αδειοδότηση. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 θα ε, μπορεί να διευρυνθεί η ευρωπαϊκή διαδικασία διοδότησης σε όλα τα προϊόντα ε, με εξαίρεση τα προϊόντα τα οποία ε, πληρούν τα κριτήρια αποκλεισμού. Όσον αφορά τα τέλη, νομίζω ότι χρειαζόμαστε σαφείς διατάξεις. Αυτό είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι κόστος θα πρέπει να φέρουν κατά την εξέταση των ουσιών η ECHA θα πρέπει ε, να ε, εισπράττει τέλεια για να μπορεί να λειτουργεί καλά. Αλλά θέλουμε να αποφύγουμε άλλες, άλλα τέλη, άλλες φορές ε, που θα εισπράττουν οι διάφοροι οργανισμοί ή τα κράτη-μέλη. Αυτό αντίκειται στην ενιαία αγορά. Χρειαζόμαστε εδώ δηλαδή ισότητα και θα πρέπει να το αποφασίσουμε αυτό σε κάποια νομοθετική πράξη κατά εξουσιοδότηση. Η αγορά βιοκτώνων είναι μικρή αγορά και γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να υπαρχει σωστή αναλογία κόστους ε, ε, όφελους. Δεν μπορεί ένας ε, παραγωγός να ζητάει την αδειοδότηση στη χώρα όπου αυτό είναι πιο οικονομικό. Επίσης, ε, έχουμε τον ε, ορισμό των ε, ευαίσθητων ομάδων. Αλλά για να υπάρχει ασφαλής χρήση των βιοκτώνων χρειάζονται κατευθυντήρες γραμμές, χρειάζεται κάποια οδηγία για την σωστή τους χρήση ώστε να προστατεύονται οι χρήστες και οι καταναλωτές και να ενημερώνονται σχετικά με τους κινδύνους. Ε, για παράδειγμα, ε, ε κάποιος που ασχολείται με παρασιτοκτόνα κτλ. θα πρέπει να ε, έχει λάβει την απαραίτητη κατάρτιση. Επίσης, στην πρώτη ανάγνωση συζητήσαμε πολύ μια διατύπωση που να αναφέρεται στους ε, κινδύνους αλλά ε, στην ε, κοινή θέση ε, αναφέρονται τα προϊόντα ε, για την παραγωγή των οποίων ε, έχουν χρησιμοποιηθεί βιοκτώνα, τα οποία όμως δεν περιέχουν τελικά βιοκτώνα. Για παράδειγμα, για την κατασκευή ενός βιβλίου έχουν χρησιμοποιηθεί βιοκτώνα, το βιβλίο όμως δεν περιέχει βιοκτώνα. Έτσι τίθεται το ερώτημα αν θα πρέπει και τα προϊόντα αυτά να εμπίπτουν στην οδηγία για, για τα βιοκτώνα. Ε, εμείς επανεισάγαμε τη διατύπωσή μας από την αρχική εκδοχή του κειμένου. Ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει ε, να καταλήξουμε σε ένα κείμενο ε, που να δείχνει ότι όλοι εννοούμε το ίδιο. Για τα ζώα και την προστασία τους έχουμε συζητήσει με την Κομισιόν και έχουμε συζητήσει ποιε είναι οι τροπολογίε οι οποίε είναι απαραίτητε και έχουμε συμφωνήσει για τα θέματα αυτά στην πρώτη ανάγνωση. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε και άλλες τροπολογίες οι οποίες θα είναι αξιόπιστες και οι οποίες θα έχουν σαν στόχο την προστασία των ζώων αλλά και οι οποίες θα έχουν και μια μορφή αυτοπεριορισμού μέσα στα πλαίσια της λογικής για τα νανοηλικά. Ήδη στην οδηγία για τις novel foods, για τα νέα τρόφιμα, έχουμε αντιμετωπίσει το θέμα αυτό το Συμβούλιο βέβαια δεν δέχτηκε αυτή την, ε, τον ορισμό τον οποίο είχαμε προτείνει. Η Κομισιόν έχει δεσμευτεί να παρουσιάσει ένα νέο ορισμό μέχρι το τέλος του χρόνου. Ελπίζω λοιπόν ότι η Κομισιόν θα μπορέσει να μας πει πότε έχει πράγματι ένα τέτοιο ορισμό και ποια μορφή έχει αυτός ο ορισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ η ίδια εκπλήσωμαι γιατί το Συμβούλιο έχει ανακατέψει με τον τρόπο αυτό τα άρθρα και πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια άλλη σειρά άρθρων αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα δεν έχουν διευκολυνθεί με το θέμα αυτό και αν διαβάσει κανείς όλη αυτή την οδηγία σαν συνολικό πακέτο θα πρέπει να μπορεί να κατανοήσει περί τίνος πρόκειται. Είναι απαραίτητο λοιπόν να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κοινή θέση του Συμβουλίου προς την κατεύθυνση αυτή και ελπίζω θα καταφέρουμε στη δεύτερη ανάγνωση να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για τα θέματα αυτά και είμαι έτοιμη να ακούσω και τις ε, παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κρίστα Κλάς για την παρουσίαση των τροπολογιών σε σχέση με τη δεύτερη ανάγνωση. έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο ήδη αντιμετωπίσαμε με τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Θα πρέπει να μείνουμε στις λύσεις των 27 κρατών μελών που είναι μεμονωμένες ή θα πρέπει να περάσουμε σε μια ευρωπαϊκή ρύθμιση. Και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει από τα κράτη-μέλη κάποια εμπιστοσύνη στις ευρωπαϊκές λύσεις και επιμένουν τα κράτη-μέλη στους δικούς του ορισμούς, τις δικές τους ρυθμίσεις για τα θέματα αυτά. Πιστεύω ότι η λογική της εσωτερικής αγοράς είναι να βρούμε ευρωπαϊκές λύσεις. Έχουμε τώρα και δύο σκιώδεις εισηγητές, είναι πολύ καλό αυτό. Ο Νταν Γιόργενσεν πρώτος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Κλά την εισηγήτριά μας. πολλά θετικά στοιχεία υπάρχουν στην έκθεσή της. και πιστεύω ότι ήταν πολύ καλή και η εισαγωγή που μας έκανε εδώ. Θα ήθελα ιδιαίτερα να την ευχαριστήσω που τόνισε την ανάγκη ε, για μια οδηγία για την βιώσιμη χρήση των βιοκτώνων. Αυτό από την αρχή ήταν πολύ σημαντικό θέμα για τη δική μου πολιτική ομάδα και χαίρομαι που όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να το πετύχουμε αυτό. Είναι μια προτεραιότητα για μας, στην οποία επιμένουμε και το Συμβούλιο θα πρέπει να το δεχτεί αυτό. Χαίρομαι επίσης για το κομμάτι που έχει να κάνει με τα πειράματα σε ζώα, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο την υποκατάσταση στον τομέα αυτό, χωρίς βέβαια αυτό να γίνεται εις βάρος της ασφάλειας. Οι σκιώδεις εισηγητές ε, κατόπιν έκκλησης της εισηγήτριας ε, έχουν κάνει πολλή δουλειά και έχουμε καταλήξει έτσι σε μία κοινή θέση ε, η οποία μπορεί να βελτιωθεί σε κάποια μέρους σημεία αλλά γενικά την στηρίζουμε. Πάντως είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε περιορισμό των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου ε, με μετατροπή των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σε εφαρμοστικές πράξεις. Ε, όσον αφορά την επιτροπολογία δηλαδή, επιμένουμε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι το Συμβούλιο πιστεύει ότι θα δεχτούμε κάτι τέτοιο. Μερικές φορές έχει κανείς την εντύπωση ότι το Συμβούλιο προτείνει κάτι το οποίο ξέρει ότι θα χάσει τελικά μόνο και μόνο για να έχει καλύτερα διαπραγματευτική θέση. Αν ε, αυτό ισχύει στην περίπτωση αυτή, εντάξει, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Ε, Τούτων λεχθέντων ε, υπάρχουν ε, ακόμα κάποιοι τομεί όπου πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες ε, τροποποιήσεις σε σχέση με τις τροποποιήσεις που πρότεινε η κυρία Κλάς. Και θα ήθελα να αναφέρω τους τομείς αυτούς, θα είμαι σύντομος. Καταρχήν όσον αφορά τα exclusion criteria, τα κριτήρια αποκλεισμού. Πιστεύουμε ότι τα κριτήρια αυτά δεν είναι αρκετά καλά, θα πρέπει να... συμπεριλάβουμε εδώ και κάποια ακόμα και επίσης όσον αφορά τις ε, εξαιρέσεις από τα κριτήρια αποκλεισμού, derogations to the exclusive criteria, αυτά οι εξαιρέσεις αυτές θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μια ε, ε, τέτοια εξαίρεση. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα δηλαδή, αλλά να είναι πολύ δύσκολο να πετύχει κανείς εξαίρεση και στην περίπτωση αυτή να υπάρχει και ένα σχέδιο υποκατάστασης. Ο άλλος βασικός τομέας έχει να κάνει με τις εθνικές ε, παρεκκλήσεις, διότι συμφωνώ απόλυτα με τον πρόεδρό μας, τον Γιώ Λάινεν, ότι ο στόχος μας εδώ είναι να έχουμε κοινή ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι σαφές ε, λοιπόν ότι όταν έχουμε ε, μια ευρωπαϊκή ρύθμιση ε, εάν δηλαδή λαμβάνεται απόφαση σε μια χώρα η οποία να ισχύει σε όλες τις χώρες ή ε, η απόφαση να λαμβάνεται σε κεντρικό σημείο μπορεί να υπάρχουν κάποιες περιστάσεις σε μια συγκεκριμένη χώρα που να σημαίνει ότι πρέπει κανείς να αρνηθεί την χρήση εμπορία αυτού του βιοκτώνου. Η κυρία Κλάση ήταν ε, ε, εισηγήτρια και όσον αφορά τα παρασιτοκτόνα ε, και θα ήθελα να πω ότι στο σημείο αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα. Και ο λόγος δεν είναι ότι δεν θέλουμε μία κοινή ευρωπαϊκή λύση. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να πετύχουμε μία κοινή ευρωπαϊκή λύση. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι τα νανοηλικά. Και εδώ πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα ξεχωριστά και θα ήθελα να ακούσω τη θέση της Κομισιόν, ε, αν και εκείνη πιστεύει ότι χρειάζεται εδώ μια ξεχωριστή προσέγγιση. Και επίσης ε, το θέμα του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα αφορά ε, μόνο τα βιοκτώνα που χρησιμοποιούνται ως βιοκτώνα ή ότι μπορεί να ε, ισχύει και για προϊόντα ε, όπου ο βασικός στόχος δεν είναι βιοκτώνος. Για παράδειγμα, κουνουπιέρες οι οποίες να έχουν επεξεργασία με βιοκτώνα. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, ε, δεν ξέρω αν έχετε προβλέψει κάτι τέτοιο. Εγώ θα ήθελα πολύ να ακούσω την ε, στάση της ε, ECHA ε, για την κοινή θέση. Βλέπω ότι είναι παρούσα η υπηρεσία αυτή. Αφού, αφού έκαναν τον κόπο να έρθουν από την Φιλανδία, νομίζω θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε τη θέση τους. Ευχαριστώ, Νταν Γιώργενσεν, η Κορίν Λεπάζ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα συμφωνήσω σε πολλά με τον κύριο Γιώργενσεν. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για όλες τις προσπάθειες, την εισηγήτρια για όλες τις προσπάθειες, αλλά λυπάμαι γιατί η ισορροπία που βρήκαμε στην πρώτη ανάγνωση απέχει αρκετά από αυτήν που, την οποία έχουμε σήμερα. Όπως είπε και ο κύριος Γιώργενσεν για την αηφορία στη χρήση δεν υπάρχει πρόβλημα για τα κριτήρια αποκλεισμού. Χρειάζεται ένα ελάχιστο. Εγώ βλέπω εδώ τις διατάξεις ε, για τους ε, ενδοκρινολογικούς ε, διαταράκτες. Στην πρώτη ανάγνωση στο 2α ορίζαμε σαφώς τι είναι ένας σήμαντος κίνδυνος. Όριζε όρια για τους ενδοκρινολογικούς διαταράκτες ε, και ε, μιλούσε για υποκατάστατα. Αυτά για τα κριτήρια αποκλεισμού. Για τις ενεργές ουσίες τώρα εγώ θα ήθελα να έχουμε τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για τις, για τις ουσίες που δημιουργούν ανώσιο τοξο, τοξικά ε, ανοσιοτοξικές παρενέργειες και νευρο, νευρολογικές διατραχές. Εγώ υποστηρίζω την κυρία Κλάς για, τις, ε, για τους ορισμούς που δίνει για τις ε, νανοτεχνολογίες. Εγώ δεν είμαι πεπισμένος, πεπισμένη ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε το Συμβούλιο. Η Κομισιόν προτείνει να αλλάξουμε τον κανονισμό για τα βιοκτώνα για να μπορέσουμε να το προσαρμόσουμε. Θα ήθελα να έχουμε επίσης και τις περιβαλλοντολογικές συνέπειες στην εφαρμοστική έκθεση και θα ήθελα να διατηρήσουμε τον κατάλογο των επιτρεπομένων ούσιων για τους μηχανισμούς χορήγησης άδειας. Για τις κοινοτικές άδειες. Εγώ πιστεύω ότι το σύστημα που προτείνει το Συμβούλιο είναι λογικό γιατί προβλέπει προοδευτικά ε, την εφαρμογή μέχρι το 2017 όπου η Κομισιόν μπορεί να εφαρμόζει την κατάσταση ανάλογα με τις ανάγκες για την απλουστευμένη άδεια. Είναι ενδιαφέρουσα αλλά η εφαρμογή αφήνει, μας δημιουργεί προβλήματα. Στο παράρτημα 1 ορίζονται τα κριτήρια για τις ουσίες που μπορούν να εγγραφούν. Πρώτο πρόβλημα, το Συμβούλιο ήδη έχει εγγράψει τις ουσίες σε αυτό το πρώτο παράρτημα 1 χωρίς να ξέρει πάνω σε ποιες βάσεις το κάνει και βάση ε, ποιων κριτηρίων. Δηλαδή τι νόημα έχει να δίνει κανείς τα προϊόντα χωρίς να έχει τα κριτήρια. Είναι περίεργο αυτό. Σύστημα αδειών για τις ουσίες και όχι μόνο για τα προϊόντα. Μα αυτό είναι κάτι το εφικτό ή όχι. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω. Περιμένω τις απαντήσεις της Κομισιόν και της εισηγήτριας σχετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λεπάζ. Προβλέπετε και μία παρέμβαση της Υπηρεσίας για τις Χημικές Ουσίες, του κύριο Μάλ, ο οποίος ήρθε από το Ελσίνκι για να μας εκφράσει την άποψη του φορέα του. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η άποψη της ΕΣΑ, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως ε, Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων από την ΕΚΑ, εγώ προετοιμα... προετοιμάσω τις ε, μελλοντικέ ενέργειες για, την... για τον κανονισμό των ε, βιοκτώνων και ο εκτελεστικός διευθυντής μου ζήτησε να τον αντικαταστήσω εξ ονόματος της ΕΤΣΑ. Η υπηρεσία μας χαίρεται πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση να συμμετάσχουμε στην συζήτηση αυτή θεωρούμε ότι είναι σημαντικές αυτές οι προετοιμασίες για μια νέα εντολή και είμαστε προσιλωμένοι στην επίτευξη υψηλής ποιότητας στο εγχείρημα αυτό. Ελπίζω ότι η εμπειρογνωμοσύνη σε τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο της ΕΚΑ θα μπορέσει να είναι πολύ χρήσιμη όπως και στην περίπτωση του REACH στις διεργασίες σας. Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για την ΕΚΑ είναι φυσικά το θέμα των ε, πόρων που συνδέονται με τα μελλοντικά καθήκοντά μας. Οι ανθρώπινοι πόροι μας είναι πραγματικά ήδη στο όριο των δυνατοτήτων τους. Η οδηγία για τα βιοκτώνα επίσης προβλέπει μια σαφή ε, διάκριση μεταξύ της χρηματοδότησης των δράσεων στο REACH και για τα βιοκτώνα και παρά το γεγονός ότι θα υπάρξουν συνέργειες μεταξύ των δύο ε, οδηγιών θα πρέπει να κρατήσουμε χωριστή τη λογιστική για τα θέματα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το, εισόδιο, το εισόδημά μας από το REACH για εγχειρήματα που έχουν να κάνουν με τα βιοκτώνα. Γι' αυτό πρέπει να υπογραμμίσω ότι οι ανάγκες σε πόρους της ΕΚΑ θα πρέπει να επανεξεταστούν μέσα στα πλαίσια ενός νέου δημοσιονομικού πλαισίου από τη στιγμή που θα έχει εγκριθεί το τελικό νομικό κείμενο. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να <clears throat> ε, δω την, ε, βλέπω θετικά την ε, ψηφοφορία της Επιτροπής σας για τα θέματα του προϋπολογισμού. Γνωρίζουμε ότι μικρές τεχνικές ε, αλλαγές σε ένα πολύπλοκο ρυθμιστικό σύστημα όπως αυτό των διοκτών μπορεί να έχει μεγάλες επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την λειτουργία της σύνολης διεργασίας αυτής. Από την άποψη αυτή εμείς χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τις τεχνικές τροπολογίες που υπέβαλε η συγγητρία που θα ευνοήσουν και την πρακτική εφαρμογή του μελλοντικού κανονισμού. Επειδή δεν υπήρξαν άμεσες ερωτήσεις προς την ΕΚΑ, εγώ θέλω να σταθώ μονάχα σε μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα για μας. Σε ό,τι αφορά το, την εμβέλεια της ευρωπαϊκής έγκρισης, εμείς φυσικά χαιρετίζουμε την διεύρυνση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της ΕΚΑ για να μπορέσει η νέα αυτή διαδικασία όμως ενωσιακής έγκρισης να επιτύχει, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, αυτό θα πρέπει να περιλάβει σαφείς διατάξεις στο νομικό κείμενο, ώστε να μην προκύψει ένα σύστημα το οποίο θα είναι υπερβολικά πεπλεγμένο. Και από τη δική μου άποψη, η πρότασή σας που μας φαίνεται ότι είναι απόλυτα λειτουργική. Κατά δεύτερο λόγο, οι πόροι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι στην ΕΚΑ για να μπορέσει να επομιστεί και το νέο αυτό έργο και να παράσχει τις νέες αυτές υπηρεσίες που τις ζητούνται και εδώ όπως είπατε μικρές αλλαγές μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους πόρους της ΕΚΑ και επομένως θα πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση των προβλέψεων για την ε, χρηματοδότηση της ΕΚΑ μετά από την έγκριση αυτού του κειμένου. Το πιο σημαντικό στο σημείο για την ενωσιακή έγκριση η, το κλειδί της επιτυχίας είναι η βαθμία διεύρυνση της ενωσιακής έγκρισης για τα διοκτώνα. Αυτό είναι μια νέα διαδικασία για ευρωπαϊκό επίπεδο και παρά το γεγονός ότι υπάρχει εθνική εμπειρία στα θέματα έγκρισης προϊόντων, αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο και γι' αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε την φάση δημιουργίας ικανότητος και μαθητείας που να μπορέσει να ακολουθήσει μια πορεία αντίστοιχη με αυτή που στην εμπειρία μας είδαμε και με το REACH όπου χρειάστηκε να υπάρχει μια σειρά φάσεων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πλήρως τα καθήκοντά μας. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει με και σταδιακό τρόπο η διεύρυνση στο, στην εμβέλεια της ενωσιακής έγκρισης και επίσης θα πρέπει να υπάρξει και σωστή καταμέτρηση του φόρτου εργασίας βάσει των προβλεπωμένων αιτήσεων για να μπορούμε να γνωρίζουμε κάπως καλύτερα τι μπορούμε να αναμένουμε. Είδαμε και την ε, συζήτηση για τα θέματα δοκιμασίας επιζώων και χαιρόμαστε για το γεγονός ότι οι κύριες αρχές, δηλαδή η αποφυγή περιττών δοκιμασιών σε ζώα, είναι ακριβώς αυτές οι οποίες περιλαμβάνονται και στην τρέχουσα πρόταση, όπως και στο REACH, και πιστεύουμε λοιπόν ότι και για τα βιοκτώνα θα πρέπει να είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε και την πολύ καλή πληροφορία και επιστημονικού χαρακτήρα που θα μπορεί να συλλέγεται για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια αυτών των βιοκτών, ενώ συγχρόνω αποφεύγονται περιττές δοκιμασίες σε ζώα. Για μας είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό και εμεί δίνουμε συνεχώς συμβουλές για τα θέματα δοκιμασιών και αυτή η εμπειρία μας ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να βοηθήσει να υπάρχει μεγαλύτερη συνέργεια με τα μελλοντικά καθήκοντά μας για τα βιοκτώνα. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ και είμαστε στη διάθεσή σας προφανώς για ό,τι περαιτέρω θα θέλατε να ρωτήσετε. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που η ECHA βλέπει θετικά την ευρωπαϊκή αδειοδότηση. Είναι περίεργο που υπάρχει ευρωπαϊκή αδειοδότηση για ε, τα χημικά, όχι όμως για τα βιοκτώνα. Αναφερθήκατε στους ε, στο θέμα των πόρων και του δυναμικού. Ε, καλέσαμε την Κομισιόν να πάρει θέση. Παρόν είναι ο Πάτρικ Μέρφυ από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Κύριε Μέρφυ, σας παρακαλώ να παρουσιάσετε τη θέση σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να τονίσω ότι το θέμα των βιοκτώνων αποτελεί προτεραιότητα για την Κομισιόν. Πρόκειται για χημικά προϊόντα για τα οποία είναι πολύ σημαντικό να αναβαθμίσουμε την νομοθεσία μας όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πιστεύουμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό από την πλευρά μας για να πετύχουμε συμφωνία κατά τη δεύτερη ανάγνωση. Σημειώνουμε με ευχαρίστηση την ε, σύγκληση που ε, έχει υπάρξει μεταξύ των διαφόρων ε, κειμένων και νομοθετημάτων το τελευταίο 18μηνο. Το τελευταίο κείμενο αποτελεί σημαντική βελτίωση της αρχικής πρότασης της Κομισιόν και πάνω από το 50% των κοινοβουλευτικών τροπολογιών υιοθετήθηκε Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει σύγκληση μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων και γι' αυτό ε, έχει βελτιωθεί σημαντικά το κείμενο. Θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο συνάδελφος από την ΕΧΑ. ότι το κείμενο αυτό αντιμετωπίζει κάποια σημαντικά πολιτικά θέματα και γεφυρώνει τις θέσεις ε, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου Υπάρχουν όμως και πολλά τεχνικά θέματα τα οποία έχουν λυθεί. Στο κείμενο των 250 σελίδων αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το κείμενο να είναι όσο πιο ε, σαφές και αποτελεσματικό διότι θα ισχύσει τα επόμενα 10 με 15 χρόνια και είναι πολύ σημαντική η σωστή εφαρμογή του κειμένου. Ε, κύριε Πρόεδρε, θα γνωρίζετε ότι η Κομισιόν ε, στα μέσα Αυγούστου υιοθέτησε ε, ανακοίνωση στις 11 Αυγούστου νομίζω, ε, η οποία έχει διαβιβαστεί πρόσφατα στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε κάποια σημεία κλειδιά, κάποια βασικά σημεία της ανακοίνωσης αυτής της Επιτροπής. Καταρχήν όσον αφορά το θέμα των πράξεων κατεξοδότηση και των εφαρμοστικών πράξεων, η Κομισιόν εφιστά την προσοχή σε δύο ε, συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, όπου κατά τη γνώμη της ε, τουλάχιστον όσον αφορά τις δραστικές ουσίες προτιμούμε τις πράξεις κατοξιδότηση και όσον αφορά τη δευτερογενή νομοθεσία για τα τέλη. Και αυτό αρχικά στην πρόταση της Κομισιόν ήταν πράξη κατοξιοδότηση, τώρα ε, ε, αναφέρεται εφαρμοστική πράξη στην περίπτωση αυτή, αλλά εμεί θα προτιμούσαμε πάλι πράξη κατοξιοδότηση. Η ε, ημερομηνία θέση σε εφαρμογή μπορεί να φαίνεται λεπτομέρεια, αλλά όπως το υπολογίζουμε εμείς, το πακέτο αυτό πιθανό είναι να τεθεί σε ισχύ, αν πετύχουμε συμφωνία κατά τη δεύτερη ανάγνωση, στα μέσα του 2012. Ωστόσο, η ημερομηνία θέση σε ισχύ ε, που αναφέρεται είναι η 1η Ιανουαρίου 2013. Ο συνάδελφος από την ΕΧΑ ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι εφαρμόσιμη η πράξη αυτή και θα γνωρίζετε ότι δεν μπορούν να δοθούν ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέχρι να ε, γίνει επίσημη υιοθέτηση του κειμένου και θέση σε ισχύ, το οποίο σημαίνει ότι η ΕΧΑ δεν θα έχει ε, πρόσβαση στις ενισχύσεις ε, του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα μέσα του 2013. Η ΕΧΑ λοιπόν χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστεί για την εφαρμογή του κειμένου και γι' αυτό στην ανακοίνωσή μας προτείνουμε η ημερομηνία θέση σε ισχύ να μεταφερθεί ε, να είναι Σεπτέμβριος του 2013 ώστε να ε, έχει η ΕΧΑ έναν χρόνο που θα, θα έχει λάβει την επιχορήγηση, θα έχει τη δυνατότητα να προσλάβει το απαραίτητο προσωπικό για να διασφαλίσει την ε, σωστή εφαρμογή του κειμένου. Μια τελική παρατήρηση που έχει να κάνει με την ανακοίνωση της Επιτροπής, ε, που έχει να κάνει με τους πόρους και το δυναμικό. Ε, κατά τις διάφορες τροποποίησεις που έχουν προταθεί στο κείμενο, η Κομισιόν πάντα έλεγε ότι ένα από τα βασικά ενδιαφέροντά μας είναι να διασφαλίσουμε το κείμενο αυτό και ο κανονισμός να μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά. Έγιναν πολλές τροποποίησεις στο κείμενο του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο εθέτησε πολλές από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, αλλά ε, το αποτέλεσμα αυτών είναι ότι ε, ε, έχει αυξηθεί πολύ ο φόρτος εργασίας για την ΕΧΑ. όσον αφορά για παράδειγμα τις ε, ε, ε, τεχνικές αντιστοιχίες, τις επιτροπές, την διαβίβαση δεδομένων και την εμπιστευτικότητα. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε εμείς στην ανακοίνωσή μας ήταν να προσθέσουμε στην ανακοίνωσή μας σε αναθεωρημένη έκδοση του οικονομικού δελτίου όπου ε, σημειώνουμε το δυναμικό που θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της η ΕΧΑ. Και αναφέρεται επίσης ε, η ευρωπαϊκή επιχορήγηση. Θα δείτε λοιπόν στο οικονομικό δελτίο ότι δίδεται περισσότερο βάρος στην αρχή όσον αφορά την ευρωπαϊκή επιδότηση, ότι θα δοθεί μεγαλύτερο μέρος της επιδότησης στην αρχή, με βαθμία μείωση μετά. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις ε, σχετικά με τις ερωτήσεις που τέθηκαν από τους ε, βουλευτές όσον αφορά τα νάνο υλικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σας λέει εδώ και αρκετό καιρό ότι ε, σύντομα θα παρουσιάσει μια ε, σχετική μελέτη. Ε, το σύντομα όμως ε, τώρα πια μάλλον σημαίνει εντός κάποιων εβδομάδων. Θα μπορέσετε να διαβάσετε λοιπόν σύντομα μία σύσταση και να κρίνετε εάν ο ορισμός που δίνεται εκεί είναι κατάλληλος και αν μπορούν να τον εγκρίνουν και τα διοθεσμικά όργανα όσον αφορά τα ε, προϊόντα που ε, έχουν υποστεί επεξεργασία με βιοκτώνα. Ε, από τότε που είδαμε το κείμενο του Συμβουλίου έχουμε ακούσει ανησυχίες από το σχετικό βιομηχανικό τομέα για τα προϊόντα αυτά. Ένα θέμα ερμηνείας είναι μήπως τα δύο θεσμικά όργανα προσπαθώντας να ε, διασφαλίσουν την σωστή ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το τι ε, περιέχουν τα διάφορα προϊόντα. Ε, εδώ υπάρχει μια ανησυχία μήπως η Κομισιόν έχει υπερβάλει και έτσι κάθε έτοιμο προϊόν που διατίθεται στην αγορά, ε, βιβλία, εφημερίδες, ε, γλάστρες, ε, θα πρέπει να, περιέχουν, θα πρέπει να έχουν την σχετική επισήμανση που να λέει ότι έχουν υποστεί επεξεργασία με βιοκτώνα κατά κάποιο στάδιο της παραγωγής. κάποια έπιπλα ε, μπορεί να ε, προκαλέσουν ε, αλλεργική αντίδραση και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν τη σχετική επισήμανση. Αλλά προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, μάλλον δημιουργήσαμε άλλα, να καταλήξουμε δηλαδή σε χιλιάδες προϊόντα τα οποία θα πρέπει να έχουν σχετική επισήμανση. Υπάρχει λοιπόν Ε, η ανάγκη να βρούμε τη σωστή ισορροπία, να φροντίσουμε οι καταναλωτές να λαμβάνουν την ε, απαραίτητη πληροφόρηση, αλλά να μην καταλήξουμε σε μια μακρά σειρά προϊόντων ε, που θα πρέπει να έχουν σχετική επισήμανση, ενώ αυτό είναι περιττό. Όσον αφορά την αηφόρο χρήση, η Κομισιόν πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνεται σωστή χρήση των βιοκτώνων. Μία από τι ανησυχίε μας είναι ότι όταν ε, βλέπουμε αυτά που θα πρέπει να κάνουν η ΕΧΑ, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη τα επόμενα πέντε χρόνια για την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, ε, δημιουργώντα ε, μια νέα διαδικασία για την αναθεώρηση των ουσιών που υπάρχουν ή για την αδειοδότηση νέων προϊόντων, νέων βιοκτώνων προϊόντων. θα πρέπει να έχουμε καμιά τριανταριά ε, δευτερογενών νομοθετικών πράξεων Και βέβαια η σωστή χρήση είναι μία από τις προτεραιότητές μας ε, για τα επόμενα 4 ή 5 χρόνια. Ε, Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό θέμα, αλλά ε, δεδομένου του φόρτου εργασία που θα έχουμε για την ε, εφαρμογή αυτής τη νομοθεσία, δεν ξέρουμε ε, αν η σωστή χρήση των βιοκτώνων βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μα. Επίση, μα απασχολεί το θέμα τη σωστή μεταχείριση των ζώων. Τη καλή μεταχείριση των ζώων. Θέλουμε να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία ε, να έχουμε προστασία των ε, καταναλωτών, προστασία του περιβάλλοντος και ε, μείωση στο ελάχιστο δυνατό των δοκιμών σε ζώα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την υπομονή σας, για το χρόνο που μου δώσατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μερφή. Και τώρα δίνω το λόγο στο Συμβούλιο, κύριε Βότσοκ, ως πρόεδρο της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου που αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά για να μας μεταλαμπατεύσει τις ιδέες που προέρχονται από αυτήν την ομάδα για τη θέση του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ε, χαιρετήσω εκ βάθους καρδίας όλους. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απαυθύνατε και για το γεγονός ότι το ζήτημα αυτό έχει ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και αποτελεί μία ακόμα από τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την συγγήτρια, την κυρία Κλάς για το γεγονός ότι ήδη έχει αντιμετωπίσει αυτό το θέμα σε ήδη πρώιμο επίπεδο και έχει αντιδράσει στην κοινή θέση του Συμβουλίου. Αυτό το θέμα είναι πολύ δύσκολο, πολύ τεχνικό και επεπλεγμένο. Δύο χρόνια δουλεύουμε στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διεργαστεί και φυσικά περιμένω θα υπάρξει περαιτέρω επεξεργασία και από τη δική μας πλευρά και για το γεγονός αυτό θα πρέπει εμείς να έχουμε τη σωστή προετοιμασία για τα επόμενα βήματα. Αυτό το οποίο δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεχάσουμε είναι ο χρόνος ο οποίος δεν περιμένει τη δική μας βραδιτήτα όπως έλεγε και ένας Πολωνός φιλόσοφος. Όλα αυτά θα πρέπει να μας οδηγήσουν να συγκεντρώσουμε περισσότερο την προσοχή μας σε αυτόν τον κανονισμό. και η Πολωνική Προεδρία είναι έτοιμη να συμβάλλει σε αυτό το στόχο. Εγώ σας ε, εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι μπόρεσα να παρασταθώ σε αυτή τη συζήτηση. Θα περιοριστώ μονάχα σε ορισμένε παρατηρήσεις που κατά την άποψή μου είναι απαραίτητο να σας δώσω την άποψη του Συμβουλίου. Μην λησμονήσετε όμως το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε ακόμα ως Προεδρία κάποια εντολή για να παρουσιάσουμε μια κοινή θέση. Μπορώ λοιπόν <clears throat> γι' αυτό το λόγο να παρουσιάσω όχι μια πλήρη θέση αλλά μονάχα ορισμένα συγκεκριμένα στοιχεία. Η κυρία Κλάς αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεκτικότητας αυτού του νομοθετήματος με άλλα νομικά κείμενα και επίσης σε ό,τι αφορά την εσωτερική συνοχή του κειμένου του Συμβουλίου. οι τεχνικές τροποποιήσεις <clears throat> που τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα και εμείς τις βλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι πολλές από αυτές τις τροπολογίες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και μπορούν να θεωρηθούν και ως χρήσιμες. Μπορούν να βελτιώσουν λοιπόν το κείμενο αυτές οι τροπολογίες. Σε ό,τι αφορά τώρα την ευρωπαϊκή ή ενωσιακή διαδικασία έγκρισης, πιστεύω ότι είναι ένα από τα κεντρικά σημεία αυτού του κανονισμού. Πιστεύουμε ότι η προσέγγιση του Συμβουλίου είναι λογική και ισορροπημένη και ότι λαμβάνει υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως από τον ε, κύριο Έχερ, μάλλον συγγνώμη τον ε, εκπρόσωπο της ΕΧΑ. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε υπόψη λοιπόν τι γνωμοδοτήσεις του φορέα αυτού της ΕΧΑ ή ΕΚΑ, που θα είναι ο φορέας ο οποίος θα επιφορτιστεί με την εφαρμογή όλων αυτών των διατάξεων που θα περιέχονται σε αυτό το έγγραφο. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και τους εκτελεστικούς κανόνες και τις πράξεις κατεξουσιοδότηση, αυτό το θέμα το έχετε τονίσει ιδιαίτερα και θα ήθελα να σας πω ότι το Συμβούλιο δεν έχει σαν στόχο να περιορίσει τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Αλλά <clears throat> όλα αυτά τα οποία έχει δεχθεί το Συμβούλιο ήταν μονάχα μετά από λεπτομερείς αναλύσεις και έχουμε ορισμένα στοιχεία τα οποία εξαρτώνται και από τον τρόπο εφαρμογής. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν μια καλή διαδικασία και επίσης και οι εθνικοί εμπειρογνώμονες θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί θα πρέπει να επηρεάσουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων Και σε ό,τι αφορά τώρα τα προϊόντα τα οποία έχουν τύχη επεξεργασίας με βιοκτώνα, αναφερθήκατε στο θέμα αυτό. Ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια λύση η οποία να είναι καλή και πρακτική και η οποία εξασφαλίζει την ασφάλεια. Και επίση πρέπει να εξασφαλίσουμε και μια ισορροπημένη λύση ό,τι αφορά την ετικετοθεσία και τη σήμανση των προϊόντων αυτών. Αυτό το τόνισε και η Κομισιόν, δεν πρέπει να το παρακάνουμε σε καμία κατεύθυνση. Για τα νανοηλικά. Νομίζω τα είπε όλα εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. <clears throat> Αναμένουμε αδειμόνως τα αποτελέσματα των εργασιών που έχουν ξεκινήσει από την Κομισιόν και κάτι ακόμα το οποίο θέλω να σας προσθέσω σε ό,τι αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξης αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε μελλοντικέ συζητήσεις αλλά θέλω να σας παραπέμψω και στο, στο παράτημα 6 που αφορά τη διαδικασία συναπόφασης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πράγματι στην πρώτη ανάγνωση είχε προτείνει ότι τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να εκχωρηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το παράτημα 6 είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του κανονισμού αυτού γιατί αφορά τις κοινέ αρχές για την τεκμηρίωση που αφορά την αξιολόγηση των βιοκτώνων σε ό,τι αφορά τη, τη δυνατότητα αηφόρου χρησιμοποίησης αυτών των διοκτώνων. Επίσης, όπως αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα ο κύριος Γιώργενσον, αυτό θα είναι και αντικείμενο περαιτέρω συζητήσεων, αλλά σε ό,τι αφορά τα ίδια αυτά τα διοκτώνα, είναι πολύ πεπλεγμενέστεροι η διαδικασία από ότι αυτή που αφορούσε προηγούμενες αντιμετωπίσεις τοξικών ή επικίνδυνων υλικών. Έχουμε 22 κατηγορίες. Θα χρειαζόμασταν μέχρι το 2020 για να αξιολογήσουμε όλες τις ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα ορισμένες ομάδες κινδύνου. Δεν έχουμε λοιπόν να κάνουμε εδώ πέρα κάτι το οποίο μπορεί να προσωμιωθεί με αυτά που κάναμε για τις επικίνδυνες και τοξικές ουσίες. Αλλά αυτό το οποίο είναι δεδομένο και σαφές είναι ότι χρειαζόμαστε να έχουμε μια λογική προσέγγιση για τα ζητήματα αυτά. Πιστεύω ότι αυτά που ανέφερα ήταν τα σημαντικότερα θέματα. Πιστεύω ότι όπως είπα και προηγουμένως, μας πιέζει ο χρόνος, τώρα είναι επικείμενη η δεύτερη ανάγνωση. Σε λίγες εβδομάδες θα πρέπει να πετύχουμε αυτά που δεν πετύχαμε στα προηγούμενα δύο χρόνια και γι' αυτό σημαίνει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στα πιο σημαντικά θέματα στη διαπραγματεύση. ευχαριστώ πολύ κύριε Βόλτσοκ, λέει ο πρόεδρος. Θα εργαστόμεν με οκίτητα Υπάρχει ο χρονικός ορίζοντας για τη δεύτερη ανάγνωση. Κρίστα Κλάς, λοιπόν. Τι θες να πεις καταληκτικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε ακόμα. Έχουμε πολλά τα οποία υποκρύπτονται ακόμα στο ευρύτερο πλαίσιο. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω ενθουσιαστεί από τον ευρωπαϊκό ενθουσιασμό με τον οποίο εμφορείται το Συμβούλιο και η Κομισιόν για να υπάρξει ένα κοινό ευρωπαϊκό εγχείρημα για τα βιοκτώνα όπως και για την φυτοϊγειονομική προστασία. Ξεκινάμε λοιπόν εδώ ουσιαστικά από την αρχή και νομίζω ότι είναι κάπως αντιφατικό να λέμε ότι θα διατηρήσουμε τις εθνικές αρμοδιότητες και μετά θα περάσουμε σε ευρωπαϊκή διαδικασία έγκρισης. Αυτό δεν βγάζει νόημα. Εγώ θα ήθελα να ακούσω από την Κομισιόν και το Συμβούλιο ότι θα ξεκινήσουμε πραγματικά προς την κατεύθυνση μιας ενωσιακής διαδικασίας, γιατί αλλιώς θα καταλήξουμε σε μια διαδικασία αμοιβαία αναγνώρισης. Αλλά σε ό,τι αφορά το αν είναι αυτό η καλύτερη λύση για την εσωτερική αγορά, εγώ πρέπει να εκφράσω τις αμφιβολίες μου. Δεν πρέπει λοιπόν να λησμονήσουμε ότι έχουν σημαντικό χαρακτήρα οι ρυθμίσεις για τα βιοκτώνα γιατί υπάρχουν και προϊόντα στην αγορά τα οποία δεν ήταν τα ίδια βιοκτώνα αλλά είχαν ένα, ένα κατά κάποιο τρόπο ένα βιοκτώνο ε, αποτέλεσμα όταν χρησιμοποιούνται σε έπιπλα, σε σκεύη, οικιακής χρήσης κτλ και διότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάποια ε, αντίδραση <clears throat> σε σχέση με αυτές τις ουσίες. Όλες αυτές τις ουσίες λοιπόν πρέπει να ληφθούν υπόψη στον ορισμό για τα βιοκτώνα προϊόντα. Εγώ άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, οι οποίοι είπαν «Ε, ναι βεβαίω να υπάρξει ενωσιακή έγκριση, ναι κύριε Γιώργενσεν. Αλλά λέτε ότι πρέπει να υπάρχουν και εξαιρέσει και για τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο οι εθνικές εξαιρέσεις να μπορέσουν να γίνουν σαφέστερες πού και πώς και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούν να υπάρχουν εθνικές εξαιρέσεις. Το ίδιο αφορά και τα κριτήρια αποκλεισμού και τα λεγόμενα σημεία αποκοπής, τα cut-offs. για τις ουσίες, τις ενεργές ουσίες οι οποίες χρήσουν αντικατάστασης θα πρέπει να είναι κάτω από μια ιδιαίτερη επιτήρηση και τότε πιστεύω θα είναι χρήσιμο να υπάρξει μια ευρωπαϊκή ταξινόμηση όλων αυτών των ουσιών. Και αυτό επί τη βάση κριτηρίων τα οποία θα είναι ποσοτικά και μετρήσιμα. Γιατί υπάρχουν πολλές ακόμα ουσίες οι οποίες δεν έχει να σαφώς καθοριστεί, δεν έχει υπάρξει συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης ή καταμέτρησή τους και ξέρουμε ότι ήδη από πειράματα σε ζώα αυτές οι ουσίες θα πρέπει να μειωθεί η χρήση τους. Όλα αυτά είναι σαφή. Υποστηρίζω την ΕΧΑ όταν λέω ότι χρειάζεται ένα νομικό κείμενο το οποίο να είναι σαφές και εφαρμόσιμο, επομένω όχι πολύπλοκο. Εργαζόμαστε προς εκεί, αλλά νομίζω ότι όσο πιο πολύ μπαίνουν στο παιχνίδι, τόσο πιο πολύπλοκο γίνεται το κείμενο. Εγώ ελπίζω ότι στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να συμπεριλάβουμε περισσότερες ουσίες. Αλλά υπάρχει και το θέμα του κόστους που θα πρέπει να υπομισθούν οι παραγωγή βιοκτώνων προϊόντων όταν θέλουν να υπάρξει η έγκριση αυτού του προϊόντος και θα πρέπει αυτό το κόστος να είναι ένα κόστος το οποίο είναι εφικτό, μπορούν να το επομισθούν. Να μην ξεχνάμε ότι οι παραγωγοί βιοκτώνων δεν έχουν μια τεράστια αγορά και τεράστια έσοδα όπως αυτοί που παράγουν φυτογειονομικά προϊόντα ή χημικά προϊόντα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια σωστή προσέγγιση για τους παραγωγούς αυτούς, αυτή είναι η ελπίδα μου, και γι' αυτό υποστηρίζω το να έχουμε δύο καταλόγους, να μιλάμε όχι για προϊόντα χαμηλού κινδύνου, αλλά για τα προϊόντα τα οποία μπορούν να περάσουν μια πιο γρήγορη και εύκολη διαδικασία έγκρισης και επομένως και σε αυτά τα προϊόντα πρέπει να είναι πιο ε, φτηνή και εποφέλης η διαδικασία από ό,τι για τα πιο επικίνδυνα προϊόντα. Είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει λοιπόν να προχωρήσουμε σε συζήτηση για τα θέματα αυτά. Τώρα βλέπω ότι δεν υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι παρόντε. Νομίζω ότι πολλά μπορούν να γίνουν με γραπτή διαδικασία και κάνω μια έκκληση προ του συνεργάτε των βουλευτών που είναι ακόμα εδώ να ζητήσουν από του βουλευτέ του να μπορέσουν να στείλουν έστω και εγγράφο τι προτάσει του ώστε να μπορέσουμε τελικά να καταλήξουμε σε ένα ε, καλό ψήφισμα γιατί όπως είπε και ο Πρόεδρός μας είναι αρκετά στενά τα χρονικά πλαίσια. Χαίρομαι λοιπόν για τις τροπολογίες και είμαι ανοιχτή για περαιτέρω συζητήσεις. Ευχαριστούμε Κρίστα. 12 Σεπτεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα είναι η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών. Ε, ψηφοφορία εδώ 4 Οκτωβρίου. Επόμενη ε, συνεδρίαση ε, στο Στρασβούργο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 και 4. Ε, κλείνουν οι συνεδρίες, θα τα πούμε τη Δευτέρα στο Στρασβούργο.